Καλημέρα κύριε και κύριοι. Παρακαλώ βάλτε τα ακουστικά σα γιατί θα μιλήσω τσεχικά. Έχουμε λοιπόν το πρόγραμμα και την ημερήσια διάταξη για σήμερα το πρωί. Έχουμε τρία πάρα πολύ ενδιαφέροντα σημεία στην ημερήσια διάταξη και θα μπορέσουμε να συνομιλήσουμε με την κυρία Τόνε Σκόγκαν, ε, υφυπουργό αμήνης της Νορβηγίας. Στη συνέχεια έχουμε θέματα ε, ασφαλείας, εξωτερικής ε, πολιτικής και έχουμε διάφορους εκπροσώπους της Ουκρανίας ε, έχουμε την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης της Ουκρανίας. Ε, ελπίζω να είμαστε στη θέση να εγκρίνουμε τη μέση διάταξη. Θα ήθελα να δώσω αμέσως το λόγο ε, στην Υφυπουργό Αμήνης της Νορβηγίας. Θέλω να σας καλωσορίσω θερμότατα στη σημερινή συνεδρίασή μας και πραγματικά εκτιμούμε το γεγονός ότι ήρθατε στην Επιτροπή μας. Θα θέλαμε να ακούσουμε την παρουσίασή σας και μετά να συζητήσουμε το θέμα των σχέσεων και ε, της πολιτικής ε, ε, κατάστασης στο Βόρειο Πόλο και στην Αρκτική γενικότερα και τις σχέσεις Νορβηγίας και Ρωσίας. Δεν είναι μέλος βέβαια η Νορβηγία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά την τελευταία δεκαετία συμμετέχει στις εργασίες που γίνονται εκεί στο Βόρειο Ατλαντικό και σε θέματα πολύ σημαντικά συμφωνούμε με την Νορβηγία γενικότερα. Υπάρχει μια συναντήληψη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και ε, θα σας δώσω το λόγο για μας κάνετε μια εισαγωγή και στη συνέχεια θα ακολουθήσει η συζήτηση. θα κάνουν ερωτήσει οι συνάδελφοι, θα απαντήσουν ή θα σχολιάσουν τα όσα είπατε και μετά θα σας παρακαλέσω και πάλι να απαντήσετε και να συνοψίσετε για να ολοκληρωθεί η συζήτηση. Ωραία. Έχουμε μία ωρίτσα περίπου μαζί σας. Παρακαλώ, έχετε το λόγο, Υπουργέ. Thank you. Uh, Ευχαριστώ πολύ και καλημέρα σας. Είναι προνόμιο για μένα που με προσκαλέσατε σε αυτήν την ε, εξέχουσα Επιτροπή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και είναι και μια πολύ καλή ευκαιρία για να μοιραστώ μαζί σας κάποιες ε, σκέψεις όσον αφορά την πολιτική μας ασφάλεια και όσον αφορά τη συνεργασία μας με την Ευρωπαϊκή Ένωση στο θέμα της ασφάλειας. Επίσης, Πρόεδρε, θα μιλήσω και για αυτά που μου ζητήσατε Θα αρχίσω λέγοντας την κοινοτυπία ότι η Νορβηγία είναι στενός συνεργάτης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμμετέχουμε στην ενιαία αγορά και για τον εξοπλισμό άμυνας και συμμετέχουμε και στην περιοχή Σέγγεν. Συνεργαζόμαστε λοιπόν για να αντιμετωπίσουμε κοινέ προκλήσεις όπως είναι η κλιματική αλλαγή, οι οικονομικές και κοινωνικές διαφορές αλλά και το μεταναστευτικό. Η Νορβηγία επίσης στηρίζει έντονα την ε, κοινή εξωτερική πολιτική και πολιτική άμυνα της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας λοιπόν προκειμένου να βελτιώσουμε τις στενές αυτές σχέσεις που έχουμε και αυτό με την ανάπτυξη μέσων που ήδη έχουμε στη διάθεσή μας αλλά και ψάχνοντας να βρούμε νέους τομείς και νέους τρόπους. Και έτσι σε λίγο θα μπω σε περισσότερες λεπτομέρειες. Όμως να σας πω και λίγα πράγματα όσον αφορά την πολιτική ασφάλειας της Νορβηγίας γενικά. Κύριος στόχος της νορβηγικής ασφάλειας και της σχετικής πολιτικής μας είναι να διασφαλίσουμε την κυριαρχία της χώρας μας, την εδαφική ακαιρεότητα και πολιτική ελευθερία δράσεων. Το πλαίσιο του διεθνούς δικαίου Ηνωμένα Έθνη, ΝΑΤΟ και διατλαντική συνεργασία στον τομέα της ασφάλειας αποτελούν και τον κρογονέο λίθο της πολιτικής μας για την ασφάλεια και την άμυνα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση επίσης είναι κάτι πολύ σημαντικό γιατί είναι το κύριο μέσο που υπάρχει για την ενότητα στην Ευρώπη και την αλληλεγγύη. Η πολιτική ασφάλεια της Νορβηγίας είναι συνδεδεμένη βέβαια με την γεωγραφική μας τοποθέτηση στην ε, βόρεια άκρη της Ευρώπης, στο βαθύ βορρά. Άρα και αυτό το θέμα είναι προτεραιότητα για μας. Υπάρχουν όλο και περισσότερες εντάσεις. Υπάρχει μια σχετική σταθερότητα στην περιοχή και ο γενικός μας στόχος είναι ακριβώς αυτή να τη διατηρήσουμε. Σταθερότητα, δηλαδή ε, βιώσιμη ανάπτυξη, διεθνή συνεργασία είναι τα κύρια στοιχεία της πολιτικής μας γενικά. Όμως βλέπουμε να υπάρχει μια νέα δυναμική και στη δικιά μας περιοχή. Κλιματική αλλαγή, για παράδειγμα, οδηγεί σε νέε ανθρώπινε δραστηριότητες στην Αρκτική, εκμετάλλευση νέων οπόρων, μεταφορές και τουρισμός. Έχουμε περισσότερες εμπορικές δραστηριότητες στην Αρκτική, λοιπόν, οι οποίες δεν θα έχουν απαραίτητα αρνητικές συνέπειες στην ασφαλεία μας. Η σύμβαση του ΟΗΕ για το δίκαιο της θάλασσας αποτελεί το πλαίσιο προκειμένου να λύσουμε τα περισσότερα θέματα που αντιμετωπίζει η περιοχή. Και οι πόροι φυσικού αερίου κλπ. αποτελούν ε, συγκεκριμένα ζητήματα κυριαρχίας στην περιοχή. Προς το παρόν δεν βλέπουμε τίποτα άλλο για την Αρκτική. Όμως, οι συνέπειες μιας Ρωσίας όλο και πιο δραστήριας είναι κάτι που μας απασχολεί. Η Αρκτική αποκτά όλο και περισσότερη σημασία για τη Ρωσία και όσον αφορά τους πόρους της αλλά και όσον αφορά το στρατιωτικό σκέλος. Η Χερσόνησος Κούλη, η οποία βρίσκεται στα σύνορα με την Νορβηγία, εξακολουθεί να αποτελεί ε, το μέρος όπου βρίσκεται η ρωσική βάση. Έχουμε τη μεγαλύτερη συγκέντρωση μη δυτικών στρατιωτικών ε, μονάδων. Επίσης, η Ρωσία έχει αλλάξει την ικανότητά της όσον αφορά την κρίση για το πώς θα συμπεριφερθεί και πώς θα ε, προχωρήσει για να αντιμετωπίσει την επικοινωνία Αμερικής-Ευρώπης. Και μέσα σε όλα αυτά βρίσκεται φυσικά και η Νορβηγία. Όλες αυτές οι εξελίξεις έχουν επιπτώσεις και στην Νορβηγία και στο ΝΑΤΟ. Ακόμα και αν δεν θεωρήσουμε την Ρωσία άμεση στρατιωτική απειλή κατά της Νορβηγίας. Μέρος της απάντησης πάντως είναι η συνέχεια οι αμυντικές δυνάμεις της Νορβηγίας που είναι ήδη ανεπτυγμένες στο βαθύ βορρά αποτελούν μια εγγύηση για την ειρήνη. Αυτή η στρατιωτική παρουσία είναι πολύ σημαντική για να διασφαλίσουμε τη συνειδητοποίηση, για να υπάρχει μόνιμη παρουσία, κυριαρχία και σταθερότητα όπως επίσης και προβλεψιμότητα. Όσον αφορά λοιπόν την ασφάλεια, πρέπει επίσης να δούμε ότι υπάρχει και ανάγκη να ενισχύσουμε την ε, εθνική μας αμυντική δύναμη. Αυτό σημαίνει να βελτιώσουμε την ετοιμότητά μας και την προμήθεια νέων στρατιωτικών εξοπλισμών, ε, μαχητικά αεροσκάφη, ε, αεροσκάφη επιθεώρησης και υποβρύχια. Και επίσης να ξαναδούμε πώς λειτουργεί ο στρατός μας. Η Νορβηγία θα βασιστεί στην ενίσχυσή μας από τους συμμάχους σε περίπτωση πολέμου και φυσικά και θέλουμε ενισχυμένη παρουσία των συμμάχων μας στο Βορρά. Φέτος το φθινόπωρο θα φιλοξενήσουμε ασκήσεις κοινέ με 35.000 συμμετέχοντες. Ο μεγαλύτερος αριθμός που συμμετέχει σε άσκηση στην Νορβηγία εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Οι δραστηριότητες αυτές ενισχύουν τη συλλογική άμυνα. Δεδομένης τώρα στη ρωσική πολιτική στην Ουκρανία. Η Νορβηγία έχει ευθυγραμμιστεί με την πολιτική κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της, ε, της στρατιωτικής συνεργασίας στα πλαίσια του ΝΑΤΟ. Συγχρόνως, στόχος μας είναι να έχουμε μια ισορροπημένη προσέγγιση. Έχουμε μακρά ιστορία συνεργασίας με την Ρωσία στο Βορρά. Συνεχίζουμε λοιπόν να συνεργαζόμαστε με την Ρωσία σε διάφορους τομείς. Αλία, για παράδειγμα, ε, συναριοφυλακή, έρευνα, ε, διάσωση και μια άμεση γραμμή στην, ε, μεταξύ Νορβηγίας και Ρωσίας. Αυτή είναι η συνεισφορά μας στην περιφερειακή σταθερότητα στο Βορρά. Δεν θα ασχοληθώ μόνο με το ΝΑΤΟ, βέβαια, στην ομιλία μου, αλλά το ΝΑΤΟ αποτελεί βασικό πυλώνα της πολιτικής ασφάλειας της Νορβηγίας. Και το ΝΑΤΟ, όπως και η Ευρωπαϊκή Ένωση, σήμερα αντιμετωπίζει σοβαρές προκλήσεις τόσο Ανατολών όσο και νοτίως. Οι εξελίξεις στο ΝΑΤΟ όμως δεν είναι κάτι που πρέπει να το δούμε ανεξάρτητα από τις εξελίξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Νορβηγία στηρίζει λοιπόν την ιδέα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να λάβει μεγαλύτερο ρόλο στην ασφάλεια και την άμυνα. Είναι απόλυτα φυσιολογικό και αναπόφευκτο. Γι' αυτό χρειάζεται συντονισμό στην Ευρωπαϊκή Ένωση που θα αναλάβει περισσότερες ευθύνες για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Είναι κάτι θετικό και για τις διατλαντικές μας σχέσεις, γιατί εκφράζει την ιδέα του επιμερισμού του βάρους. Συνεπώς, τα τελευταία 20 χρόνια η Νορβηγία είχε ως στόχο τη συνεργασία αυτή εν ώψη τέτοιων εξελίξεων στην Ευρώπη. Για την εξωτερική μας πολιτική, για παράδειγμα, έχουμε παράδοση να ευθυγραμμιζόμαστε στις δηλώσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα περιοριστικά μέτρα. Έχουμε συνεισφέρει και εμείς στη διαχείριση πολλών κρίσεων και συνεισφέρουμε σημαντικά στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Άμυνας. Παρακολουθούμε επίσης με ιδιαίτερο ενδιαφέρον τις πιο πρόσφατες πρωτοβουλίες που ξεκίνησαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ενισχυθεί περισσότερο η ΕΠΑ. Χρειάζεται περισσότερο σχεδιασμό, ικανότητα, ε, μόνιμες δομές συνεργασίες και η δημιουργία ενός αμυντικού ταμείου. Η Νορβηγία επίσης συμμετέχει ως μόνη χώρα μη μέλος στην έρευνα ΠΕΣΚΟ τώρα, η EDF και η ΕΠΑ όλα είναι ευπρόσδεκτα. Είναι όμως πολύ σημαντικό να βαθύνουμε περισσότερο στις πολιτικές αυτές, χωρίς όμως να δημιουργηθούν νέες διαχωριστικές γραμμές στην πολιτική ασφάλειας. Και έτσι έρχομαι στο επόμενο θέμα μου, που είναι η συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Μετά την κοινή δήλωση της Βαρσοβίας, έχει επιτευχθεί σημαντική πρόοδο στη συνεργασία μεταξύ των ε, δύο πλευρών. Τώρα αναγνωρίζεται σαφώς ότι αντιμετωπίζουμε τις ίδιες προκλήσεις όλοι. Οι πόροι ανήκουν στις ίδιες χώρες μέλη. Το θέμα λοιπόν δεν είναι πώς να αποφύγουμε μόνο επικαλύψεις, ε, αλλά πώς θα διασφαλίσουμε τη λειτουργικότητα. Ο νέος δυναμισμός της ESDP που συνδυάζεται με την σημερινή κατάσταση ασφάλειας αποτελεί και σημαντικό κίνητρο για να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ των δύο πλευρών. Έχουμε πολλές προτάσεις έτοιμες για τέτοια συνεργασία. πώς θα υλοποιηθούν όλα αυτά. Αυτή είναι η πρόκληση. Γι' αυτό στόχος μας πρέπει να είναι να προχωρήσουμε σε ένα περιορισμένο αριθμό προτάσεων κοινού ενδιαφέροντος. Και το πιο ενδιαφέρον είναι να μειώσουμε τα εμπόδια στην ε, μετακίνηση στρατιωτικών δυνάμεων στα ευρωπαϊκά σύνορα σε περίπτωση κρίσης ή πολέμου. Είναι κάτι που πρέπει να μπορούμε να πετύχουμε μέχρι τη διάσκεψη του Ιουλίου και έτσι να έχουμε μια νέα κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Υπάρχει περιθώριο επίσης για περισσότερη συνεργασία και στα Δυτικά Βαλκάνια. Για ασκήσεις. Οι σχέσεις ΝΑΤΟ-Ευρωπαϊκής Ένωσης αποτελούν στοιχείο κλειδί για την ε, επερχόμενη διάσκεψη του ΝΑΤΟ και άρα πρέπει να έχουμε αυτά αποτελέσματα εκεί. Επιτρέψτε μου επίσης να πω και δύο λόγια για το Brexit δημιουργείται ένας νέος δυναμισμός στην ε, συνεργασία για την άμυνα συγχρόνως με το Brexit. Το Brexit βοήθησε να ε, απελευθερώσει τις ικανότητές της η Ευρώπη. Αυτό είναι κάτι ήδη πολύ σημαντικό. Από πλευράς Νορβηγίας είναι ζωτική σημασίας να διασφαλίσουμε ότι θα υπάρξει ένας νέος δυναμισμός στην ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άμυνας χωρίς αρνητικές συνέπειες στις άλλες πλευρές, Ευρωπαϊκή Ένωση, Ηνωμένο Βασίλειο, Νορβηγία για παράδειγμα. Πρέπει να αποφύγουμε αποδυνάμωση της πολιτικής μας αυτής μετά το Brexit. Συγχρόνως όμως θέλουμε το Ηνωμένο Βασίλειο να διατηρήσει ένα ρόλο ως σημαντικός παίχτης στην πολιτική αυτή και την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Τα πιο πρόσφατα δείγματα που έχουμε από το Ηνωμένο Βασίλειο δείχνουν ότι θέλει να συμμετέχει πλήρως στην ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Και αυτό είναι βέβαια ευπρόσδεκτο. Συγχρόνως όμως γνωρίζουμε ότι οι διευθετήσει συμμετοχής του Ηνωμένου Βασιλείου ξεπερνούν αυτά τα οποία έχει η Νορβηγία σήμερα. Η σε διευθετήσεις λοιπόν για την πολιτική αυτή είναι κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολύ και την Νορβηγία. Η Νορβηγία δεν συμμετέχει στις διαπραγματεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ηνωμένου Βασιλείου, αλλά μας ενδιαφέρει και έχουμε απόλυτα θεμητό συμφέρον να ξέρουμε τι γίνεται, ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Γιατί είναι κάτι που έχει να κάνει με τη στενή μας συνεργασία της Καλλιώς σε πολλούς τομείς και εσωτερικών, αλλά και σε σχέση με την δικιά μας τη συμμετοχή στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας. Συνεπώς, θέλουμε να υπάρξει συνεχής διάλογος με την Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατάσταση πραγμάτων στις διαπραγματεύσεις αυτές με τον Ηνωμένο Βασίλειο. Και έτσι φτάνω και στο τελευταίο μου θέμα, που είναι η συμμετοχή της Νορβηγίας ως εταίρος στην Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας. Είναι πολύ σημαντικό η πολιτική αυτή να αναπτύσσεται με διαφάνεια και με δυνατότητα για τους συμμετέχοντες και τους ε, συμμάχους που δεν αποτελούν μέρος της. Όπως ε, είπαμε, η Νορβηγία ενδιαφέρεται όλος ιδιαιτέρως, για όλος έχουν ε, να κάνουμε την Ευρωπαϊκή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας. Και αυτό έχει να κάνει με τη συμμετοχή μας αυτή όλα αυτά τα χρόνια που είχαμε συμμετάσχει σε τρεις στρατιωτικές και νέες μη στρατιωτικές αποστολές. Και επίσης έχουμε δυνάμεις και στη, στα πεδία μάχης της Ευρώπης. Έχουμε στους μάχημους δηλαδή σχηματισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Συμμετέχουμε λοιπόν στην πολιτική αυτή, παρόλο που δεν είμαστε χώρα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τέλος, οκτιμούμε όλους ιδιαίτερως τις δυνατότητες που δίνονται σε τρίτες πλευρές να συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση στην ασφάλεια και την άμυνα. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν περιθώρια παρετέρω βελτίωση σε διάφορους τομείς κλειδί. Ιδιαίτερα. Περισσότερη συμμετοχή σε συζητήσεις, διαμόρφωση αποφάσεων, και ενημέρωση. Είναι κάτι το οποίο θα βοηθούσε τη συμμετοχή και θα βοηθούσε την συνεισφορά μας στην πολιτική ασφάλειας και άμυνας να γίνει ακόμα πιο ελκυστική. Πιστεύουμε ότι μια τέτοια συμμετοχή μπορεί να επιτευχθεί καλύτερα με διαφοροποίηση μεταξύ των διαφέρων χωρών εταίρων, λαμβάνοντας υπόψη τα χαρακτηριστικά της κάθε χώρας, του κάθε εταίρου δηλαδή να είναι περισσότερο à η προσέγγιση. Για την Νορβηγία είναι πολύ σημαντικό να μας προσκαλείτε να συμμετέχουμε και στο δεύτερο στάδιο της EDF και κυρίως σε διάφορα προγράμματα. Η συμμετοχή μας εδώ θα ήταν προς όφελος όλων των πλευρών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα αυτό και για πολλούς λόγους. Πρώτα όλα, η αμυντική βιομηχανία της Νορβηγίας είναι εχμής και ανταγωνιστική διεθνώς και παίζει σημαντικό ρόλο στην ε, αλυσίδα της ευρωπαϊκής αμυντικής βιομηχανίας. Δεύτερον, για την Ευρωπαϊκή Ένωση η Νορβηγία είναι ένα σημαντικό εταίρος γιατί συμμετέχει πλήρως στην αγορά αμυντικού εξοπλισμού της Ευρώπης και συνεργάζεται όσον αφορά τον εξοπλισμό και είναι και σημαντικός πελάτης της ευρωπαϊκής ε, αμυντικής βιομηχανίας. Και θα ήταν περίεργο να μειώσουμε την ε, συμμετοχή αυτή, δεδομένου που συμμετέχουμε πλήρως και στην εσωτερική αγορά. Συνεπώς, όλες οι χώρες έχουν να αποφεληθούν. Τρίτον, μέσω της συμμετοχής μας στην έρευνα. Η νορβηγική αμυντική βιομηχανία θα συνεισφέρει σημαντικά στην έρευνα όσον αφορά τις αμυντικές ικανότητες. Πρέπει να συμμετέχουμε στην έρευνα, στις αμυντικές ικανότητες, και να μην αποκλειόμεθα βέβαια από την ανάπτυξη των ικανοτήτων αυτών. Δεν θα ήταν λογικό κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και πιστεύουμε ότι είναι αμοιβαίο το όφελος να προσκαλείται η Νορβηγία και να συμμετέχει στα προγράμματα τα αμυντικά. Με την συμμετοχή της Νορβηγίας πιστεύουμε ότι προωθείται και συνεργασία με τις χώρες μέλη και η Νορβηγία θα αναλάβει το κόστος της συμμετοχής αυτής βέβαια όσο την αφορά. Επίσης θέλουμε να έχουμε τη δυνατότητα για μελλοντική συμμετοχή και σε ε, μεμονωμένα προγράμματα ΠΕΣΚΟ. Η αμυντική βιομηχανιακή ΠΕΣΚΟ είναι ένα γενικότερο πλαίσιο. Σήμερα και η Σουδία έχει πει ότι θέλει τέτοιες ευκαιρίες συμμετοχής και συνεργασίας και εκτεταμένη συμμετοχή σε διάφορες ε, αποφάσεις επιχειρήσεων. Δυστυχώς η υπάρχει μια ε, συμμετρία όσον αφορά την Σουηδία, τη Φιλανδία και την Νορβηγία. Δεδομένου ότι το ΝΑΤΟ και η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι στρατηγική εταίροι, θα έπρεπε να θέλουμε άνοιγμα και συμμετοχή όλων των χωρών Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ. Χαιρόμαστε που η Ευρωπαϊκή Ένωση ξεκίνησε μια νέα στρατηγική προσέγγιση για τις χώρες εταίρους και ελπίζουμε ότι η διαδικασία αυτή θα αντιμετωπίζει και τις ανησυχίες που έχουν ορισμένες χώρες εταίροι όπως είναι η Νορβηγία. Το γεγονός ότι υπάρχει περιθώριο για βελτίωση δεν σημαίνει ότι πρέπει να ξεχάσουμε το βασικό μου μήνυμα που είναι ότι η Νορβηγία εκτιμάει όλους ιδιαίτερο τη δυνατότητα που έχει να συμμετέχει στενά στην, ε, στις διαδικασίες ΚΕΠΑ και έχουμε συνεισφέρει πάρα πολύ στην συνεργασία αυτή και εμείς και σαφής μας στόχος είναι να συνεχίσουμε τη συνεργασία αυτή τα επόμενα χρόνια. Είναι προς όφελος όλων των ευρωπαϊκών χωρών. Σας ευχαριστώ λοιπόν και πάλι που με προσκαλέσατε και σας ευχαριστώ και για την προσοχή σας. Ε, ευχαριστώ πολύ κυρία Υπουργέ για την παρουσίαση αυτή. Πολύ ενδιαφέρουσα. Περιγράψατε την κατάσταση ε, πάρα πολύ ε, παραστατικά και περιστατωμένα. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον κύριο Γκάλερ από το Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Ευχαριστώ πολύ. Καλώς ορίσατε θερμά, κυρία Υπουργέ, στα νορβηγικά ο κύριος Γκάλερ και σας ευχαριστώ για όλη αυτή την επισκόπηση που μας δώσατε για τη θέση της Νορβηγίας εντός του ΝΑΤΟ και βεβαίως ε, και στα πλαίσια ε, της ήδη υφιστάμενης συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Καθώς επίσης και για την προθυμία σας να συνεχίσετε τη συνεργασία αυτή και να την αναβαθμίσετε ακόμη περισσότερο. Βεβαίως είστε στην ενιαία αγορά και θα παραμείνετε. Και μπορείτε να δώσετε και το καλό παράδειγμα στο απερχόμενο κράτος μέλος για το πώς θα παραμείνει στη συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Πριν από 15 μέρες είχαμε πάει στη Φιλανδία και ρωτήσαμε ποιες είναι οι σχέσεις σας με το ΝΑΤΟ και ήταν πολύ ενθαρρυντικά αυτά που ακούσαμε. Είναι βέβαια κράτος μέλος Ευρωπαϊκής Ένωσης και όχι του ΝΑΤΟ η Φιλανδία. Είναι πολύ ενδιαφέρον και πολύ ενθαρρυντικό. Και επίση πολύ ενθαρρυντικό είναι και το αντίστροφο να είστε μέλο του ΝΑΤΟ αλλά όχι τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Πλην όμω συμμετέχετε σε όλα αυτά, στον Ευρωπαϊκό Αμυντικό Οργανισμό, τα απαριθμίσατε. Και στα υπόλοιπα, ε, στο ερευνητικό πρόγραμμα για το Ταμείο και επίση είστε πρόθυμοι να αναβαθμίσετε ε, ε, τη συμμετοχή σας στο e IDP. Ε, τώρα είμαστε στο στάδιο της νομοθεσίας και έχουμε βρει τρόπο να συμμετέχουν και τρίτες χώρες, εκτάκτος βέβαια. Αυτό φορά τη Βρετανία που στο μέλλον δεν θα είναι στην αγορά. Εσείς θα παραμείνετε στην εσωτερική αγορά, δεν είναι η δική σας περίπτωση αυτή. Υπάρχουν περισσότερες δυνατότητες για σας. Βεβαίως δεν θα πρέπει να υπάρχουν ε, νομικοί περιορισμοί ε, για το αποτέλεσμα αυτής της συνεργασίας, δηλαδή να είμαστε απολύτως κυρίαρχοι και ε, της συνεργασίας και της κατάστασης. Κάτι άλλο θέλω να ρωτήσω τώρα. Um, Πώς θα σφυριλατήσετε την απαραίτητη αντοχή και ανθεκτικότητα απέναντι στις προκλήσεις της Ρωσίας. Πριν από λίγα χρόνια είχατε αυτή την εισβολή με τα ποδήλατα, για να τη χαρακτηρίσω έτσι, με κάποιους πρόσφυγες που τους μετέφερε η Ρωσία πολύ βόρεια για να σας δείξει ε, και ε, σε εσά και στη Φιλανδία. Κοιτάξτε τι μπορούμε να κάνουμε αν θέλουμε να σας πειράξουμε λίγο και να σας τσιγκλίσουμε. Ε, εσείς πώς ε, προετοιμάζεστε και ποια είναι η σημερινή σας προετοιμασία απέναντι σε τέτοιες κινήσεις της Ρωσίας. Such Αν θέλει να επαναλάβει τέτοια επεισόδια ή ε, παρόμοια. Για την Αρκτική είπατε ότι δεν υπάρχει κούρσα για την Αρκτική για τις οικονομικές δραστηριότητες αλλά και για την ασφάλεια. Αλλά εμείς ακούμε τα τελευταία δύο-τρία χρόνια ότι η Ρωσία οργιάζει εκεί. Ε, είναι πάρα πολύ παρούσα και έχει επανενεργοποιήσει ε, παλιούς σταθμούς ε, πολύ στο, στο βαθύ βορρά και στις ακτές της και ακόμα πιο βόρεια. Εσείς πώς το βλέπετε αυτό, αυτές τις δραστηριότητε και την έντονη κινητικότητα της Ρωσίας. Αυτές τις ερωτήσεις έχω προς το παρόν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γκάλερ. Η κυρία Μούντι. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Θέλω να σας ενδια... Ε, ευχαριστήσω και εγώ για την ενδιαφέρουσα παρουσίαση. Τι να συμφωνήσω με τον συνάδελφο κύριο Γκάλερ για τα διδάγματα που θα μπορούσε να αντλήσει από εσά η δική μου χώρα, ε, το Ηνωμένο Βασίλειο, στις σχέσεις μας. Γιατί από ό,τι φαίνεται προς το παρόν την παρούσα σχέση τη διαλύουμε. σε σχέση με τα όσα είπατε για την Ευρωπαϊκή Ένωση ε, και τη συνεργασία με τον ΝΑΤΟ, πώς είναι οι σχέσεις μας, πώς ε, διαμορφώνονται, πώς θα μπορούσαμε να τις κάνουμε πιο αποτελεσματικές στο μέλλον. Ένας από τους τομείς που καλύπτεται από τη συνεργασία αυτή και φαίνεται ότι λειτουργεί καλύτερα είναι η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και ε, στην άμυνα. Εσείς ασχολείστε με το συγκεκριμένο και με ποιον τρόπο και πώς αποδίδει. Και μπορούμε να αντλήσουμε κάποια μαθήματα και από εκεί και κάποια συμπεράσματα για να βελτιώσουμε τη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ. Εσείς πώς το βλέπετε από την σκοπιά της Νορβηγίας. Και αναπόφευκτα φυσικά θέσατε το θέμα του Brexit και τις προσπάθειες που έχουν γίνει. Ποιος ξέρει τις μελλοντικές σχέσεις και τις προθέσεις της ε, κυβέρνησης Μεγάλης Βρετανίας για τη συμμετοχή στην ΕΠΑ. Εσείς, αν κατάλαβα καλά, θέλετε να συμμετέχετε. Είναι δηλωμένη σας πρόθεση αυτή να μπείτε σε αυτό το σχήμα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας. Και συμφωνώ και με τον συνάδελφο Γκάλερ για το EDIDP, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης ε, στον τομέα της άμυνας και πώς ε, συνεργάζεται με το Αμυντικό Ταμείο. Θέλετε λοιπόν να έχουμε σχέσεις πιο στενές και πιο ε, εντατικές, αλλά ε, σωστά σας κατάλαβα ότι αν υπάρχει κάποια πολύ στενή σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση θα μπορούσε να προταθεί και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν ξέρω αν ισχύει για τη σχέση που έχετε εσείς σήμερα με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αν αυτό μπορεί να μεταφερθεί και να ισχύσει και για ε, τις σχέσεις της Νορβηγίας με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βανόρτα. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να ευχαριστήσω την ε, Υφυπουργό της παρατηρήσεις Χαίρομαι που τελικά ανέφερε και το θέμα του ΝΑΤΟ. που είναι ακρογωνίως λίθος σε θέματα άμυνας και για την Νορβηγία όπως και για τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως, μιλήσατε για τον Brexit. Εσείς είστε ε, στην ενιαία εσωτερική αγορά, έχετε επίση κάτι να πει τα θέματα τα, με τα σύνορα. Ξέρουμε τα τελευταία 20 χρόνια πόσο έχει στην Νορβηγία και βεβαίως σωστά προσδίδεται μεγάλη σημασία στην προστασία της κυριαρχίας της χώρας σας. Αλλά υπάρχει και ένα μέρος το οποίο έχετε ε, επίσης Βεβαίω πάντα πρέπει κανείς να υπολογίζει σε τους καταστάσεις και τα υπέρ και τα κατά. Δεν ε, συμφωνώ με τον ενθουσιασμό σε την ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άμυνας. Αλλά βεβαίως εφόσον την έχουμε θα πρέπει με αυτήν να προχωρήσουμε. Δυστυχώς έτσι έχουν τα πράγματα. Η πραγματικότητα όμως είναι ότι αν μπορούσαμε να γυρίσουμε τα ρολόγια πίσω, κανένας δεν θα δημιουργούσε αυτή την πολιτική έτσι όπως είναι. Και πολύ σωστά είπατε ότι δεν θα πρέπει να ζούμε γύρω από διαχωριστικές γραμμές, διότι ο κύριος στόχος αυτής της ευρωπαϊκής πολιτικής ήταν ίσως να δημιουργήσει κάποιες γραμμές, γιατί μιλούσε για ε, ε, στρατηγική ανεξαρτησία και, και αυτονομία. Και έτσι καταλαβαίνουμε εμείς τα πράγματα και στο ΝΑΤΟ και λαμβάνοντα υπόψη και τι, ποια είναι η πολιτική των ΗΠΑ. Βεβαίως, θα ήθελα να σας να ζητήσω και κάτι άλλο. Αναφέρατε τη Ρωσία. Για την Κίνα, τι έχετε να πείτε. Αρχίζετε να βλέπετε με το άνοιγμα της, ε, του διάβλου αυτού του βόρειο-ανατολικού, βορειοδυτικού θέματα στην Επίσης, με τους γειτονές σας, με την Σουηδία, με τη Φιλανδία, ιδιαιτέρως. Πώς έχει το θέμα αυτό, διότι Ποτέ δεν κατάλαβα γιατί είναι εκτός ΝΑΤΟ. Θεωρούνται ότι είναι ε, στρατιωτικά ουδέτερες χώρες. Αλλά αυτή τη στιγμή ε, συμφωνούν με την ΠΕΣΚΟ, με αυτή την περίφημη ενισχυμένη ε, ε, συνεργασία. Είναι όμως εκτός ΝΑΤΟ. Και ποια είναι η θέση σας. Τι κάνετε ίσως για να τις ενθαρρύνετε να γίνουν μέλη του ΝΑΤΟ. Ευχαριστώ. Κύριε Βαν Όρντεν, η κυρία Λέζινγκ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Πολλές από τις ερωτήσεις που είχατε τις απαντήσατε ήδη. Έχω μόνο πολύ συγκεκριμένες τώρα, συμπληρωματικές και διευκρινιστικές ερωτήσεις. Αν κατάλαβα καλά, ε, το πρόγραμμα για την αποτροπή ε, συμβάντων και επεισοδίων στη θάλασσα ήταν αυτό που αναφέρεται. Και θέλω να σας ρωτήσω, τι άποψη έχετε ε, για την πρόταση του European Leadership Council να διευρυνθεί αυτό σε όλα τα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ και να δημιουργηθεί και μία συνιστόσα για τον εναέριο χώρο. Και δεύτερη συγκεκριμένη ερώτηση Διάβασα μερικές εκθέσεις και αναφορές που λένε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείες στέλνουν άρματα μάχης, πυροβολικό, ε, σε ε, προκεχωρημένες θέσεις στα σύνορα με την ε, Ρωσία για να αποκρούσουν ενδεχόμενη εισβολή. Αυτά ισχύουν που διάβασα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Λέζινγκ. Και τώρα αν μου επιτρέπετε, κυρίες και κύριοι, θέλω να κάνω κι εγώ μια ερώτηση στην κυρία Υφυπουργό. Κύριε Υπουργέ, είπατε ότι δεν θεωρείτε τη Ρωσία άμεση απειλή. Μα υπάρχουν χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση που τη θεωρούν και την παραθεωρούν άμεση απειλή. Και η Τσεχική Δημοκρατία και η Πολωνία και άλλες χώρες. Αυτό έχει να κάνει με την εγκατάσταση ε, πυράβλων ε, στρατηγικών στο Καλίνιγκραντ. Δεν υπάρχει αντίστοιχη απειλή για σας. Τι γίνεται με τις βάσεις στη Χερσόνησο Κόλα. Ε, τα ελέγχετε αυτά. Δηλαδή γνωρίζετε τι συμβαίνει εκεί, τι βαλιστικούς πυράβλους έχουν με, μετατοπίσει και τι σταθμεύει εκεί, γιατί είναι στα άμεσα σύνορά σας. Πιτέρα, Πιτέρα. Ε, κυρία Πιτέρα. <laughs> Dziękuję bardzo. Ε, ja chciałabym nawiązać do wstępu. Mm, e, θα ήθελα να σας ρωτήσω κάτι ε, για μια λευκή βίβλο που ε, δημοσιεύσατε. Ε, αφορά αυτό την εξωτερική πολιτική της Κίνας. Λοιπόν, τι γίνεται με την Κίνα. Η Κίνα προσβλέπει στη συνεργασία ε, και για τις μεταφορές ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για την εναέρια κυκλοφορία. Ε, δηλαδή, είναι πάρα πολύ έντονη η παρουσία της και το ενδιαφέρον της για τις μεταφορές. Και αυτό τώρα αφορά και τη μείωση των χρόνων που χρειάζονται για τις μεταφορές, για τις μεταφορές εμπορευμάτων με τις νέες οδούς που ανοίγουν ε, στο βορρά. Οπότε η Κίνα ενδιαφέρεται ιδιαίτερα και για τους φυσικούς πόρους και για τα κοιτάσματα που θέλει να εκμεταλλευτεί και αυτή, φυσικό αέριο κλπ. Πώς αξιολογείται αυτές τις ε, προσδοκίες και τις φιλοδοξίες της Κίνας είναι αντικείμενο συζήτησης. Θεωρείται ενδεχόμενη απειλή κάτι τέτοιο. Ε, όλα αυτά από ε, το, το, βόρειο δρόμο του μεταξιού, ας πούμε, πώς θέλουν να το χαρακτηρίσουν. Possibly elaborate on your very brief mention, you very briefly mentioned of the possible negatives in relation to the development of Θα ήθελα πάρα πολύ ε, σύντομα να αναφέρω στα πλαίσια της ευρωπαϊκής ε, κοινή πολιτικής ε, άμυνας και σε σχέση με τον Brexit πιστεύω ότι συνεισφέρει πάρα πολύ ε, το ΝΑΤΟ, κυρίως το βόρειο, με, οι δυνάμεις που βρίσκονται στο βόρειο ε, μέτωπο. Αυτό είναι κάτι το οποίο σε σχέση με την Αρκτική και την πολιτική σας έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Σε σχέση με τις συζητήσεις που γίνονται ε, επίσης για... but scant uh, Arctic warfare capability, which of course will be of importance and interest to Norwegian interests. Thank you. Ευχαριστούμε πολύ. Κύριε Υπουργέ, θα ήθελα λίγο να επανέλθω σε ένα θέμα τεχνολογίας που αναφέρατε. Η Ευρώπη δεν είναι η ηγέτης παντού στην αμυντική βιομηχανία και εδώ μιλώ για τον εξοπλισμό και του ΝΑΤΟ και τις αμυντικές ικανότητες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχουν δύο τομείς τεχνολογίας που κατά την άποψή μου είναι ε, συμπληρωματικά και αφορούν και την Νορβηγία. Ε, προβλέπετε να εξυγχρονίσετε την αεράμινά σας. Ε, γνωρίζω και θυμίζω ότι τώρα βασίζεστε ε, στο αμερικανικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών. Ε, οι Αμερικανοί όμως τώρα αναπτύσσουν νέα τεχνολογία, έχουν περάσει την επόμενη γενιά. Ε, με εσάς, τι γίνεται στην Νορβηγία. Δεύτερον, η Νορβηγία κάποτε είχε πάρα πολλά υποβρύχια και θυμάμαι πάρα πολύ καλά ότι μειώσατε το στόλο στο μισό, το στόλο των υποβρυχίων. Τώρα έχουμε νέα γενιά υποβρυχίων που αγοράζουν τα διάφορα κράτη-μέλη και ε, ε, στη ε, γερμανικά υποβρύχια κυρίως. Πώς βλέπετε τον εξυγχρονισμό του στόλου των υποβρυχίων της Νορβηγίας. Ευχαριστούμε πολύ. Δεν βλέπω να υπάρχει άλλη ερώτηση. Οπότε, κύριε Υφυπουργέ, έχετε 15 λεπτά να απαντήσετε στις ερωτήσεις αυτές. Παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα προσπαθήσω να απαντήσω με τον καλύτερο δυνατό τρόπο και να σχολιάσω τα πάρα πολύ επίκαιρα οξυδερκή σχόλια και ερωτήσεις που τέθηκαν. Πόσο βλέπω σας ενδιαφέρει πάρα πολύ η σχέση με τη Ρωσία. Πράγμα το οποίο ήταν, εάν θυμάμαι καλά, και το αντικείμενο της πρώτης ερώτησης του κύριο Ντάλλερ. Όπως προσπάθησα να πω, έχουμε μακρά παράδοση στις γειτονικές σχέσεις μας αυτές με την Ρωσία. Και Πρώτα απ' όλα θέλουμε αφενός να έχουμε καλές σχέσεις, δεδομένου ότι είμαστε γειτονικέ χώρες, έχουμε καθημερινή συνεργασία, ένθεν και ένθεν, έχουμε πολύ καλή συνεργασία στην αλληλεία και πιστεύω ότι είναι πολύ σωστός ο τρόπος με τον οποίο χειριζόμαστε το όλο θέμα των αλλιευτικών αποθεμάτων μεταξύ Ρωσίας και Νορβηγίας. Επίσης είπα ότι σε θέματα διάσωσης συνεργαζόμαστε σωστά επίσης. Τούτου λεχθέντος, ο στόχος μας είναι να είμαστε ένα ανοιχτό βιβλίο, να είμαστε ανοιχτοί και προβλέψιμοι γείτονες, να ξέρουν οι άλλοι πώς είμαστε σε διοικητικό επίπεδο πολλές φορές στο Υπουργείο Άμυνας κάνουμε συζητήσεις, ενημερώνουμε, τους ενημερώνουμε για τις επόμενες ασκήσεις, για την πολιτική μας γενικότερα, διότι πιστεύουμε ότι όταν έχουμε μία ανοιχτή και σωστή ενημέρωση, θα θεωρηθεί ότι έχουμε μία θετική στάση και συνεισφορά σε όλη την πολιτική μας. Βεβαίως, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι είμαστε άμεσος γείτονας σε ε, μία χώρα η οποία μονίμως αναβαθμίζει τον εξοπλισμό της. Ξέρουμε ότι υπάρχουν ε, πολλές δραστηριότητες, ότι υπάρχει πολύ μεγάλη ικανότητα, πολλές δυνατότητες. Πρέπει να το έχουμε αυτό κατά νου και να το αντιμετωπίζουμε. Γι' αυτό το λόγο η πολιτική αποτροπής και το γεγονός ότι εμείς είμαστε πολύ ισχυρό μέλος του ΝΑΤΟ και της Συμμαχίας είναι σημαντική. Αυτά λοιπόν αν θέλετε είναι τα δύο σκέλη της προσέγγισης μας ώστε να ισοσκελίζουμε πάντα την ε, σχέση μας με την ε, Ρωσία. Αυτό το γεγονός που αναφέρατε με τα ποδήλατα πρέπει να πω ότι είχε μεγάλο σχέση με το μεταναστευτικό ε, κύμα στο τέλος του 2015. Αλλά και πάλι μπορέσαμε να συζητήσουμε, να διαπραγματευτούμε και να καταλήξουμε για να χειριστούμε τέτοιου είδους καταστάσεις και πάλι μαζί τους. Και πολύ καλό παράδειγμα είναι το ότι πραγματικά μπορούμε και να έχουμε και με τον, μεταξύ των δύο λαών πολύ καλή σχέση. Ξέρουμε ότι είναι πιο δραστήριοι οι Ρώσοι και προσπαθούμε πάντα να συνειδητοποιούμε ότι πρόκειται για μια κατάσταση στην οποία πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και όταν βλέπουμε ότι ενισχύει, αναβαθμίζει το βόρειο μέτωπο το ΝΑΤΟ, το κατανοούμε και ησυχάζουμε. Τώρα, η ασφάλεια του κυβερνοχώρου, ε, που ανέφερε και η Ναι, θα μπορούσαμε να μιλήσουμε και μία, για μία υβριδική διάσταση. Πρόκειται για συμπληρωματικά λοιπόν στοιχεία σε σχέση με αυτά τα οποία γνωρίζαμε πολύ καλά στο παρελθόν. Αυτή λοιπόν η ασφάλεια στον κυβερνοχώρο μας κάνει να πούμε ότι όντως θα πρέπει να το αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα, ώστε να δημιουργήσουμε νέες και ισχυρές πολιτικές. Δεν θα πρέπει να θεωρούμε δεδομένο πλέον ότι όταν θα αρχίσει μια τέτοια κατάσταση να αντιμετωπίσουμε, πρέπει να δούμε πώς ε, αρχίζει μια τέτοια κατάσταση για να ξέρουμε εκ των προτέρων προ, να την αντιμετωπίσουμε. Δεν ξέρουμε πόσο θα διαρκέσει. Πρόκειται επίσης ε, για κάτι το οποίο πάντα έχει έναν άγνωστο χ πίσω από μια τέτοια είδους επίθεση. Πάντα λοιπόν θα πρέπει να εστιάζουμε περισσότερο την προσοχή μας σε όλο τον ευρύτερο τομέα της ασφάλειας στον κυβερνό χώρο. Και αυτό είναι κάτι το οποίο και η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ θα πρέπει να εξετάσουν, να μελετήσουν και να είμαστε συντονισμένοι και ευθυγραμμισμένοι στο τι κάνουμε για να αντιμετωπίσουμε τέτοιου είδους επιθέσεις. Για να δω τις σημειώσει μου. Με ρωτήσατε αν ε, η Νορβηγία θέλει να δημιουργήσει στενότερη σχέση και με να ακόμη και μετά την έξοδο της Μεγάλης Βρετανίας σε θέματα ασφαλείας και άμυνας. Πιστεύω ότι ναι, μπορούμε να βρούμε περαιτέρω τομείς, θα πρέπει να δούμε πώς οι διάφορες πρωτοβουλίες θα μελετηθούν και βεβαίως όλα αυτά εξαρτώνται από την ιδιαιτερότητα της κάθε χώρας και ο καθένας επειδή είναι διαφορετικός μπορεί να έχει τη δική του συνεισφορά. Η εσωτερική αγορά υποχωρείται κάπως σε θέματα συνόρων. Πρέπει να κάνουμε ίσως μία διαφοροποίηση μεταξύ του τι σημαίνει να είναι κανείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση εντός Ευρωπαϊκή, ε, αγοράς και τι σημαίνει για μία μικρή χώρα σαν και εμάς. Ε, εποφελούμεθα από το γεγονός ότι όντως υπάρχουν και άλλες ευρωπαϊκές χώρες και πολίτες της, της Ευρωπαϊκής Ένωσης από την αγορά εργασίας τη δική μας. Έρχονται, ε, εργάζονται και αυτό είναι εποφελές αμοιβαίως. Πιστεύω λοιπόν ότι είναι διαφορετικό το θέμα για τους εργαζόμενους από αυτό της αντιμετώπισης των, του μεταναστευτικού. Νομίζω ότι εδώ είμαστε πιο κοντά με αυτά τα οποία κάνει, τρόπο με το οποίο ενεργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και νομίζω ότι όντως είμαστε επιτυχείς στο ότι στον τομέα αυτό έχουμε μία πιο αυστηρή αλλά θετική, επιτυχή πολιτική. Όσον αφορά την Κίνα και τον και η Νορβηγία, όπως πολλές άλλες χώρες, πιστεύουν ότι υπάρχουν εξελίξεις στην Κίνα, γίνεται όλο και περισσότερο η Κίνα ένας διεθνής παίκτη και αυτό είναι κάτι το οποίο ε, παγκοσμίως μας επηρεάζει όλους. Τώρα, η Αρκτική ε, η τήξη των πάγων, η κλιματική αλλαγή μας οδηγεί στο να δημιουργήσουμε νέες ε, οδούς μεταφορών, ανάπτυξη τουριστικών δυνανοτήτων και η Κίνα επίσης ενδιαφέρεται για αυτό του είδους τα θέματα. Είπα ότι δεν θεωρούμε ότι η Ρωσία είναι απειλή και δεν πιστεύουμε ότι υπάρχει κίνδυνος ή θα υπάρξει κίνδυνος άμεσα ότι η Ρωσία θα είναι επικίνδυνη. Βεβαίως δεν μπορούμε να αποκλείσουμε το γεγονός ότι αν συμβεί κάτι τέτοιο σε μια άλλη περιοχή του κόσμου θα επηρεαστεί η κατάσταση της ασφαλείας ακόμη και σε μας, διότι όπως ελέγχθη από κάποιους το γεγονός ότι οι Ρώσοι έχουν αυτά που έχουν και κατέχουν στο βορρά, ίσως θα υπάρχει ε, αυτή η μετακύληση του προβλήματος, αν υπάρχει κάποια διαταραχή που μπορεί να φτάσει και μέχρι εμάς. Τώρα, ε, μία από τις τελευταίες παρατηρήσεις. Η παρουσία των Ηνωμένων Πολιτειών στην Νορβηγία. Όχι μόνο τον είπα, αλλά και πολλών άλλων συμμάχων, οι οποίοι είναι τα τελευταία χρόνια παρόντες. Για την ε, κατάρτιση, για τις ασκήσεις από κοινού με τα δικά μας τα στρατεύματα. Αυτό είναι σημαντικό για μας και αυτό είναι μέρος της συμμετοχής μας στον, στην ε, Βορειοατλαντική Συμμαχία διότι αναμένουμε οι σύμμαχοί μας να έρθουν να μας βοηθήσουν αν παραστεί ανάγκη. Άρα θα πρέπει να έχουν εξοικειωθεί με το κλίμα μας, με την ε, ε, γεωγραφική μας ιδιομορφία και ίσως υπάρξει μια τέτοια ε, πιθανότητα. Άρα εδώ και πάρα πολύ καιρό χαιρετίζουμε οποιαδήποτε ε, διαδραστική τέτοιου τύπου δραστηριότητα από κοινού με τους συμμάχους. Και η πολιτική μας είναι να μην έχουμε μονίμως παρουσία συμμάχων. Βρίσκονται λοιπόν ε, εκ περιτροπής για κάποια προγράμματα για να αποκτήσουν εμπειρία, αλλά όχι συνεχώς. Επίσης βλέπουμε ότι σφαιρικά έχει και μεγαλύτερη παρουσία στις ΣΥΠΑ η και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό το χαιρετίζουμε, διότι πιστεύουμε ότι πρόκειται για ένα θετικό μήνυμα το οποίο εκπέμπουν οι ΕΠΑ. Και είναι μέρος της πολιτικής τους να έχουν ισχυρά παρουσία στην Ευρώπη. Τελευταία παρατήρηση και ελπίζω ότι απάντησα σε όλα τα ερωτήματα. Η αναβάθμιση. Για τα υποβρύχια, όντως, έχουμε ένα ειδικό πρόγραμμα σε σχέση και με τη Γερμανία. Όχι μόνο αναβαθμίζουμε τα υποβρύχια, αλλά εξυγχρονούμε και την αεράμινά μας. Αγοράζουμε νέα F-35, ε, κάνουμε επισκόπηση των συστημάτων που χρησιμοποιεί ε, ο χρησιμοποιούν τα στρατεύματά μας ώστε να βελτιώσουμε το σύστημα άμυνας που έχουμε. Επίσης έχουμε αυξήσει σημαντικά σε ποστό 25% τα κονδύλια του προϋπολογισμού που ε, αφορούν την άμυνα από το 2012-2013 και ένθεν. Και κυρίως για να εξυγχρονίσουμε τον εξοπλισμό μας για τις νέες τεχνολογίες, όντως θεωρούμε ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό ε, θέμα για να ολοκληρώσουμε την μακροπρόθεσμη στρατηγική μας σε θέματα άμυνας. Ευχαριστώ, ελπίζω ότι απάντησα σε όλες τις ερωτήσεις που τέθηκαν. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Υφυπουργέ. Για δύο πράγματα κυρίως σας ευχαριστούμε. Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστούμε επειδή αντέξατε 15 λεφτά που σας δώσαμε, καταφέρατε να μας απαντήσετε. Και δεύτερον, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα όσα τόσο ξεκάθαρα και σαφή μας είπατε ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε και να περάσουμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία και υλοποίησή της. Ευχαριστώ κύριε και κύριοι. Καλημέρα σας. Um, Έχω τη χαρά και την τιμή να αναλαμβάνω την Προεδρία για την παρούσα ενότητα. Ε, καλημέρα αγαπητοί συνάδελφοι. περάσουμε στο σημείο 10 της μερίσιας διάταξης, η εφαρμογή της ΠΕΣΚΟ, της μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας. Να αρχίσω από κάτι, αν μου επιτρέπετε, που ήταν απρόοπτο. Όταν πήγαμε στην Ουάσιγκτον την περασμένη εβδομάδα με αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η πρώτη προτεραιότητα ποια ήταν στις συζητήσεις μας με τους συναδέλφους και στην Βουλή των Αντιπροσωπών και στη Γερουσία ε, για την ε, διατραντική συνεργασία. Αυτό που τους ενδιαφέρει ήταν η Πέσχο. Και ε, έπρεπε να πείσουμε και τους ομολόγους μας στο Κογκρέσο και την κυβέρνηση ότι η ΠΕΣΚΟ είναι πολύ σημαντικό όχι μόνο για τη στρατηγική ασφάλειας και άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά ότι είναι και με το ΝΑΤΟ κτλ. Πάντως αυτό που έχει ενδιαφέρον, το βασικό επιχείρημα, για να μην είναι και αυτό αντικείμενο σύγκρουσης, ήταν ότι μέχρι στιγμής δεν έχει και καμιά μεγάλη ουσία, ε, ούτε και ουσία στην σύγκρουσή μας. Η ΠΕΣΚΟ όμως η συνεργασία αυτή, η μόνιμη διαρθρωμένη, είναι από τις σημαντικότερες πρωτοβουλίες για την ασφάλεια και την άμυνα και επιταχύνεται από ό,τι φαίνεται. Έχουμε λοιπόν την ιδιαίτερη χαρά και τη μείωση και το πρενόμιο να ανταλλάξουμε απόψεις με τον αντιστράτηγο Έσα Πούλκινεν, Γενικό Διευθυντή ε, του Στρατιωτικού Επιτελείου της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τον ε, Χόρχε Ντομέκ, ε, διευθύνων ε, σύμβουλο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Εχθές ε, το Κοινοβούλιο ψήφισε ε, για ένα από τα δύο φιλόδοξα ερευνητικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την ανάπτυξη ικανοτήτων και δόθηκε και ισχυρή εντολή από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Καλωσορίζω τους ομιλητές μας. Σας ευχαριστώ πολύ που ήρθατε ξανά στην Επιτροπή και θα ήθελα να δώσω το λόγο στο μου. Συμφωνείτε, στρατηγέ. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Σας ευχαριστώ ε, πάρα πολύ για τα θερμά σας λόγια. Κάνω μια ε, δήλωση ε, γνωστή από κάποια τηλεοπτική σειρά. Έρχεται χειμώνα, μάλλον. Και στη χώρα μου αρχίζουμε να μετράμε τις θερμοκρασίες ως χειμερινές όταν κατέβει κάτω του μείον 20. Δεν έχουμε φτάσει ακόμα εκεί ε, τις επόμενες μέρες ίσως. Σε σχέση με τα όσα είπατε για τις επαφές σας με την Αμερικανική κυβέρνηση και τη διοίκηση και εγώ έχω την ίδια ε, εντύπωση αποκομίσει πριν από λίγες εβδομάδες ήμουν εκεί και η Πέσκο τους ενδιαφέρε σφόδρα να μάθουν τι ακριβώς γίνεται, περί τίνος πρόκειται και ε, θέλησαν πολύ να το συζητήσουν. Πολύ αυθεντικό και γνήσιο ενδιαφέρον έδειξαν. Ο Χόρχε γνωρίζει πολύ καλά τι είναι Πέσκο, όπως και εγώ, ότι προσπαθούμε να θεσμοθετήσουμε ε, τη συνεργασία μας ε, με, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στο ΝΑΤΟ, στη Βόρεια Ευρώπη, η Σκανδιναβία και η ε, ΠΕΣΚΟ είναι ένας διάβλος για να γίνει αυτό, να γίνει μια τυποποιημένη, ε, διαρθρωμένη συνεργασία και μόνιμη. Και αυτή είναι η βασική διαφορά με το προηγούμενο διάστημα που δεν είχαμε αυτή την πολιτική και αυτή τη συνεργασία. Θα δούμε μέχρι πού μπορούμε να εμβαθύνουμε και να διευρύνουμε. Καλή σας μέρα και πάλι. Um, Uh, Θα ήθελα να θυμίσω την απόφαση του Συμβουλίου στις 11 12 του 2017 ίδρυε τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία ΠΕΣΚΟ με 25 κράτη-μέλη που υπέγραψαν μια διακήρυξη για κοινή δέσμευση. Ε, τώρα βλέπω ότι βρισκόμαστε ε, στην αρχή μιας μόνιμης διαδικασίας. Έχει γεννηθεί η ΠΕΣΚΟ και αρχίσαμε τη διαδικασία ακριβώς ε, της ε, επιχειρησιακής της ε, λειτουργίας. Υπάρχει μια σύσταση για την εφαρμογή και μια λίστα έργων και με τα κράτη-μέλη που συμμετέχουν. Αυτές είναι αποφάσεις του Συμβουλίου που τώρα ετοιμάζονται να εγκριθούν στις 6 Μαρτίου στο Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων που θα λάβει χώρα εδώ στις Βρυξέλλες. Βεβαίως υποστηρίζουμε κρίσιμους τομείς για την ε, ΠΕΣΚΟ. Θα πρέπει να υπάρχει ένας μηχανισμός αξιολόγησης, αξιόπιστος, φιλόδοξα σχέδια και υλοποίηση φυσικά των δεσμεύσεων. Έρχομαι πρώτο στο μηχανισμό αξιολόγησης. Τι σημαίνει αυτό. Θα πρέπει να εκπονούνται ε, εθνικά προγράμματα ισχυρά και εφαρμόσιμα ε, που θα επιτρέπουν στα κράτη-μέλη να υλοποιούν τις κοινέ δεσμεύσεις. Υπάρχει το άρθρο 3 της απόφασης που ορίζει ότι τα συμμετέχοντα κράτη-μέλη εντός των εθνικών προγραμμάτων τους θα εξηγούν πώς θα φτάσουν σε αυτούς τους δεσμευτικούς στόχους και θα διευκρινίζουν ε, τους πιο συγκεκριμένους στόχους που θα θέτουν σε κάθε ε, φάση της μόνιμης διαφρομένης συνεργασίας και πώς όλα αυτά θα υλοποιούνται. Τα εθνικά αυτά ε, σχέδια θα είναι συμπληρωματικά το ένα προς το άλλο και θα ενημερώνεται πάντα το Συμβούλιο για τους στρατηγικούς στόχους ΠΕΣΚΟ. θα πρέπει να υλοποιηθούν οι δεσμεύσει. Βεβαίω το επιχειρησιακό σκέλο ακόμα δεν έχει υλοποιηθεί. Θα πρέπει να λαμβάνουν συγκεκριμένα μέτρα για τη διαθεσιμότητα, την διαλειτουργικότητα, την ευελιξία και την ανάπτυξη ε, των δυνάμεων. Ενδεχομένως μπορεί να ε, αναθεωρείται και η εθνική νομοθεσία ή να χρειάζεται κάτι τέτοιο. Η διαθεσιμότητα και η δυνατότητα ανάπτυξης των ενόπλων δυνάμεων, η διαλειτουργικότητα και η πιο φιλόδοξη δράση συνδέεται και με την κοινή χρηματοδότηση των αποστολών ΕΠΑ. Ένα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι τα φιλόδοξα σχέδια της ΠΕΣΚΟ. Το Νοέμβριο αργότερα κατά τη διάρκεια του έτους θα υπάρξει και ένας δεύτερος κατάλογος σχεδίων και η Γραμματεία ΠΕΣΚΟ ε, συμμετέχει και βοηθάει τα κράτη-μέλη στην αξιολόγηση, στη συνεργασία και ε, στην εδραίωση των διαφόρων σχεδίων. Τον Απρίλιο-Μάιο θα ήταν σκόπιμο να ε, προκηρυχθεί και η δεύτερη φάση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για σχέδια στη Γραμματεία και η Στρατιωτική Επιτροπή με τις ε, συμβούλους μπορούν να βοηθήσουν τα κράτη-μέλη για να ε, χαράσουν τα σχέδια, τα προγράμματα. Και πάλι έχουμε μια εμπειρία από την πρώτη φάση των προγραμμάτων, μια πιο διαθρωμένη ε, προσέγγιση θα ακολουθηθεί στο μέλλον, έτσι ώστε να αναπτύσσονται τα σχέδια με βάση προτεραιότητες που έχουμε εντοπίσει ε, από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας και μετά από τη συντονισμένη ετήσια αναθεώρηση ε, της άμυνας. Αυτή η πιο διαρθρωμένη λοιπόν διαδικασία θα γίνει βάση ε, κοινώς συμφωνηθέντων σχεδίων στάνταρ για να βοηθούμε τα κράτη-μέλη να κάνουν τις προτάσεις τους, τα συμμετέχοντα. Προβλέπεται σε δεύτερη φάση να συμπεριληφθούν εκτός από τα νέα σχέδια και τις προτάσεις των κρατών μελών και κάποια από την πρώτη φάση που δεν έχουν ακόμα συμπεριληφθεί. Ε, κυρίως εστιάζουμε στην ικανότητα και δεύτερον στις επιχειρησιακές προτεραιότητες. Για την επόμενη ε, προοπτική θα πρέπει να δούμε ποιες είναι οι συνέργειες και πώς συνδυάζονται ε, οι διάφορες προτεραιότητες στην ανάπτυξη στρατιωτικών ικανοτήτων και στη διεθνή συνεργασία. Πέσχο. και στο Ευρωπαϊκό Ταμείο για την Άμυνα και προς την κατεύθυνση αυτή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο πρωταγωνιστικό, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά ε, το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Βιομηχανικής Ανάπτυξης στον τομέα της άμυνας, το EDIDP, που θα συνεισφέρει πάρα πολύ όχι μόνο για τη βιομηχανία, αλλά και ε, για να αναπτύξουμε τις στρατιωτικές μας φιλοδοξίες και αυτό είναι πιο σημαντικό για μένα. Υπάρχει και μια παγκόσμια στρατηγική για την Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαι πεπισμένος ότι οι συλλογικές μας ε, προσπάθειες μέσω πρόθεσμα θα αποδώσουν ε, και θα αυξήσουν την στρατηγική αυτονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ολοκληρώνω εδώ και σταματώ. Είναι τα εισαγωγικά μου σχόλια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, στρατηγέ. Και μια που αναφερθήκατε στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, νομίζω θα πρέπει να ακούσουμε τώρα και τον επικεφαλής, τον κύριο Ντομέκ. Έχετε το λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ για την πρόσκλησή σας και την ευκαιρία που μου δίνετε να ενημερώσω την υποπιτροπή σας για την υλοποίηση της ΠΕΣΚΟ. Θέλω να αρχίσω ευχαριστώντας το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το οποίο συνεχώς ζητά την υλοποίηση των διατάξεων της Λισαβόνας όσον αφορά την πολιτική ασφάλειας άμυνας και την ΠΕΣΚΟ. 11 Δεκεμβρίου 2017, 25 χώρες μέλη ε, νόμιμα δεσμεύτηκαν υπέρ της αμυντικής ολοκλήρωσης και δεσμεύτηκαν για 20 πράγματα όσον αφορά την λειτουργικότητα και τις επιχειρήσεις. Επίσης συμφώνησαν για έναν κατάλογο 17 προγραμμάτων που θα αναλυθούν υπό την ΠΕΣΚΟ. Πρόκειται για κατάρτιση, για στρατιωτική μετακίνηση, ε, ετοιμότητα επιχειρησιακά κλπ. Η ΠΕΣΚΟ λοιπόν είναι μια διαδικασία από τις χώρες μέλη. Οπότε είναι πολύ σημαντικό οι χώρες που συμμετέχουν να αναλαμβάνουν δεσμεύσεις. Επίσης να γίνεται μια καλή αξιολόγηση και ενημέρωση των διαφόρων εθνικών σχεδίων. Τώρα πια πρέπει να αναλάβουμε και βήματα για να υπάρχει μια καλή ισορροπία ανάμεσα στην ποιότητα της εργασίας μας και την ταχύτητα υλοποίησης. Την επόμενη εβδομάδα για πρώτη φορά από τότε που ξεκίνησε η ΠΕΣΚΟ, οι Υπουργοί Άμυνας θα συναντηθούν ε, στα πλαίσια του, του Συμβουλίου Εξωτερικών υπό τη μορφή ακριβώς αυτή της ΠΕΣΚΟ. Υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου, οποία επισημοποιεί την ε, συμφωνία για διάφορα προγράμματα και ορίζει τα μέλη και υπάρχει και η σύσταση του Συμβουλίου για χάρτη πορείας όσον αφορά την υλοποίηση της ΠΕΣΚΟ. Το πρώτο βασίζεται στη δήλωση ε, των ε, μελών ε, ΠΕΣΚΟ. Όλες οι προτάσεις προγραμμάτων επιλέχθηκαν από τις χώρες μέλη τη χρονιά που μας πέρασε και αξιολογήθηκαν βάσει συγκεκριμένη μεθοδολογίας που έχει αναπτύξει ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας και η Γραμματεία της ΠΕΣΚΟ που προσφέρει η ικανότητα ε, για τα προγράμματα αυτά σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, λαμβάνοντας ε, υπόψη το πρόγραμμα ανάπτυξης ικανοτήτων και βέβαια ως κάτι συμβατό με τον ΝΑΤΟ. Οπότε υπάρχει διαμεσολόβηση και η μεθοδολογία αναπτύχθηκε με τρόπο που ικανοποίησε όλες τις χώρες μέλη. Επιτρέψτε μου τώρα να σας παρουσιάσω τα πρώτα 17 προγράμματα που επέλεξαν οι χώρες μέλη που συμμετέχουν, που μπήκαν σε τρεις κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία προγραμμάτων έχουν να κάνουν κοινέ ασκήσεις και κατάρτιση. Είναι κάτι πολύ σημαντικό και υπάρχει εδώ πέρα το στοιχείο της ανάπτυξης ικανοτήτων για να προετοιμαστούν οι δυνάμεις για επιχειρήσεις και αποστολές. Υπό το πνεύμα αυτό τα δύο πρώτα προγράμματα ε, το πρώτο για το κέντρο κατάρτισης και το δεύτερο για την πιστοποίηση της κατάρτισης όσον αφορά τον Ευρωπαϊκό Στρατό, θα προσφέρει περισσότερη συνέπεια και καλύτερη αμοιβαία κατανόηση, κατανόηση και καλύτερες ικανότητες σε όλα τα επίπεδα. Η δεύτερη κατηγορία που είναι κοινέ ικανότητες περιλαμβάνει έξι προγράμματα τα οποία θα έχουν σημαντικές επιπτώσεις στην ε, συνέπεια στην Ευρώπη και θα υπάρξει περισσότερη συνεργασία. Θα διευκολύνουν τις ε, δυνάμεις και τις διάφορες μονάδες των χωρών μελών προκειμένου να μπορούν να δημιουργήσουν μεγαλύτερους σχηματισμούς δύο προγράμματα εφαρμόζονται στις ικανότητες αυτές που βελτιώνουν την ικανότητά μας να διαχειριζόμαστε μονάδες σε μεγάλη απόσταση και να τις στηρίζουμε καλύτερα. Άλλα προγράμματα στην κατηγορία αυτή έχουν να κάνουν με την υλικοτεχνική στήριξη που είναι κάτι απαραίτητο για κάθε αποστολή και επιχείρηση κυρίως για τις μονάδες αυτές που αναπτύσσονται σε μεγάλη απόσταση. Επίσης χρειάζεται μια ροή απρόσκοπτη για στήριξη. Αυτό σημαίνει ότι χρειάζεται και αποτελεσματική οργάνωση και της ιατρικής στήριξης των δυνάμεων αυτών. Χρειάζονται βελτιωμένες διαδικασίες και ρυθμίσεις για να γίνεται πιο εύκολη μετακίνηση των δυνάμεων. Χρειάζεται επίσης ε, περισσότερη συνοχή στην Ευρώπη και κάλυψη των ε, αδυναμιών, κάτι το οποίο θα γίνει με τέσσερα προγράμματα τα οποία αλληλοσυμπληρώνονται μεταξύ τους. Πρόκειται για το ιατρικό σκέλος, πρόκειται για το δίκτυο το υλικοτεχνικό με ευρωπαϊκούς κόμβους και πρόκειται και για το πρόγραμμα ενέργειας για επιχειρήσεις. Η τρίτη κατηγορία με νέα προγράμματα περιλαμβάνει τέσσερις επιχειρησικούς ε, τομείς που έχουν να κάνουν ε, με από αέρα, θάλασσα, χερσαία κλπ. Πρόκειται για ικανότητες που έχουν να κάνουν ε, με τους επιχειρησιακούς κλάδους για να βελτιωθεί η συνοχή των ικανοτήτων στην Ευρώπη και έχουν ξεκινήσει τέσσερα προγράμματα για το χερσαίο σκέλος με στόχο να βελτιωθούν οι μάχημες ικανότητες και να εξυγχρονιστούν με νέα στοιχεία, κυρίως για το πεζικό και το πυροβολικό. Επίσης, προκειμένου να μπορούμε να ανταποκριθούμε σε περιπτώσεις καταστροφών. Τα αποτελέσματα θα τα έχουμε μέσω του προγράμματος για το πεζικό με την ανάπτυξη του πακέτου για την ανακούφιση από κρίσεις και καταστροφές. Τώρα, υπάρχει και πληροφορική. Προκειμένου να διασφαλίσουμε την επικοινωνία, πρέπει να διασφαλίσουμε τον κυβερνοχώρο. Και για να τα καταφέρουμε αυτά υπάρχουν τρία προγράμματα για τον κυβερνοχώρο και την ε, θάλασσα. Έχουμε διάφορα μέτρα για την προστασία. Η πλατφόρμα για τον κυβερνοχώρο, πρώτα απ' όλα, χρησιμοποιεί την ίδια μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για τα πρώτα προγράμματα και θα χρησιμοποιηθεί για οποιαδήποτε προτάσεις επιπλέον προγραμμάτων πέρα από τον κατάλογο που έχουμε ήδη και θα αποτελέσει μέρος του δεύτερου κύματος προγραμμάτων που θα έχουμε φέτος. Η γραμματεία ΠΕΣΚΟ θα είναι έτοιμη να συνεχίσει να στηρίζει τις χώρες που συμμετέχουν στην αξιολόγηση και στην παγίωση των προτάσεων. Επιπλέον, η γραμματεία ΠΕΣΚΟ φέτος το Μάρτιο θα δημιουργήσει ένα ενιαίο mailbox προκειμένου να υπάρχει πρόσβαση των χωρών μελών σε όλες τις υπηρεσίες. Η ΠΕΣΚΟ δεν είναι μόνο ένας κατάλογος προγραμμάτων. Η συμμετοχή στην ΠΕΣΚΟ έρχεται πρώτα απ' όλα με ισχυρή πολιτική βούληση, η οποία δείχνει την αποφασιστικότητα της χώρας να περάσει σε πιο δεσμευτικές ε, δράσεις προκειμένου να υπάρξει παρατέρω ανάπτυξη ικανοτήτων και μεγαλύτερη ικανότητα επιχειρήσεων. Όσον αφορά την υλοποίηση, η γραμματεία της ΠΕΣΚΟ προτείνει να οργανωθεί με δύο συναντήσεις του Συμβουλίου κάθε χρόνο. Απρίλιο-Μάιο, για παράδειγμα, φέτος, όπου οι Υπουργοί θα συζητήσουν την ετήσια έκθεση αξιολόγησης που τους υποβάλλει το HR το Μάρτιο η αξιολόγηση θα βασιστεί στα εθνικά προγράμματα εφαρμογής των χωρών που συμμετέχουν και που υποβάλλουν το Δεκέμβριο κάθε χρόνο οι αρχές Ιανουαρίου όπου θα αναφέρουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί την προηγούμενη χρονιά και θα περιγράφουν και τα σχέδιά τους για την επόμενη χρονιά. Τον Νοέμβριο οι Υπουργοί θα επικεντρώνονται κυρίως σε νέα προγράμματα. Προηγουμένως, από τον Απρίλιο-Μάιο μέχρι τον Νοέμβριο θα μπορούν οι χώρες να προτείνουν στη γραμματεία ΠΕΣΚΟ νέα προγράμματα. Και αυτό πριν να υπάρχουν οι στρατιωτικές συμβουλές από το ΓΙΤΟΣΥ που θα συμφωνεί με αυτές το Συμβούλιο. Αυτή είναι μια διαδοχή γεγονότων και κάθε δεύτερο χρόνο θα υπάρχει έκθεση που θα βοηθάει ε, την ενημέρωση για νέες ευκαιρίες που υπάρχουν και που θα μπορούσε να λάβει υπόψη της η ΠΕΣΚΟ. Οι χώρες μέλη συμφωνούν με προτεραιότητες και έτσι θα τροφοδοτούν την ΠΕΣΚΟ. Στα πλαίσια αυτά θέλω να αναφέρω επίσης ότι το Μάρτιο η γραμματεία ΠΕΣΚΟ θα δώσει το πρώτο της feedback όσον αφορά τις πληροφορίες που έχουν προσφέρει χώρες μέλη για τα εθνικά τους σχέδια και τι θα έχουν ανακοινώσει δηλαδή το Δεκέμβριο οι διάφορες χώρες, προκειμένου να υπάρξει συνειδητοποίηση για το είδος και για τη δομή των πληροφοριών που δίνονται από τις χώρες μέλη, έτσι ώστε στο μέλλον να μπορεί να γίνεται μια πιο ουσιώδης αξιολόγηση και προκειμένου ενημερώνονται οι χώρες που συμμετέχουν στην ΠΕΣΚΟ για να προσφέρουν πιο συγκεκριμένους στόχους και να βοηθούν στην συνέχεια των προτάσεων για προγράμματα μέχρι τον επόμενο Δεκέμβριο. Πριν τελειώσω, επιτρέψτε μου να πω και δύο λόγια για την συνολική συνοχή των διαφόρων πρωτοβουλειών. Υπάρχει η ΚΑΡΤ, υπάρχει ΠΕΣΚΟ, υπάρχει Ευρωπαϊκός Οργανισμός Άμυνας Πιστεύω ότι όπως συνεχίζουμε με την εξέλιξη όλων αυτών των πρωτοβουλειών, πρέπει να εμπεδοθούν μέσα σε μια συνολική προσέγγιση, η οποία θα πρέπει να καλύπτει από τις κοινέ προτεραιότητες μέχρι τα αποτελέσματα και τις επιπτώσεις, όπως είναι το πουλ ευρωπαϊκών δυνάμεων, και για τις ικανότητες και για τη δυνατότητα ανάπτυξης κλπ. Συνεπώς, το σχέδιο που θα έρθει τώρα τον ε, Ιούνιο θα αποτελέσει τη βάση για ενημέρωση και του Ευρωπαϊκού Ταμείου Άμυνας και των προγραμμάτων ΠΕΣΚΟ. Οι προτεραιότητες ε, επίσης της κοινή πολιτικής ασφάλειας και άμυνας θα ληφθούν υπόψη και η συνοχή με κάθε σχεδιασμό και με εθνικά σχέδια. Αποτελεί στοιχείο αναφοράς στην Ευρώπη για να διασφαλίσουμε ότι προσφέρουμε τις κατάλληλες ικανότητες και στο μέλλον. Πιστεύω λοιπόν ότι εφόσον κάνουν προσπάθειες οι χώρες μέλη που συμμετέχουν για περισσότερο δεσμευτική συμμετοχή σε προγράμματα, η ΠΕΣΚΟ θα αποτελέσει ένα πολύ βασικό στοιχείο που θα ενισχύσει τις ευρωπαϊκές δυνάμεις και θα προσφέρει μια περισσότερη συνοχή στη δράση τους. Ευχαριστώ κύριε Ντομέκ. Ο κύριος Κίλαμ είναι ο πρώτος συνάδελφος της Ταϊτολόγια. Ευχαριστώ πολύ για αυτό το ενθαρρυντικό μήνυμα. Νομίζω ότι ο σχεδιασμός είναι πάρα πολύ πιστικός και εντυπωσιακό. Όντως, η ΠΕΣΚΟ αποτελεί την ευκαιρία να ενισχύσουμε τη συνεργασία μεταξύ ε, χωρών μελών του ΝΑΤΟ και μη μελών του ΝΑΤΟ. Πριν από δύο εβδομάδες πήγαμε στην Φιλανδία και η εξαιρετική ετοιμότητα που υπήρχε για όλα αυτά και η εμπειρία των Φιλανδών μας εξέπληξε. Τώρα δεν θα πρέπει να χάσουμε αυτή την δυναμική που έχει δημιουργηθεί. Ωραία είναι λοιπόν τα σχέδια, αλλά όπως δείχνει και η πρακτική, η εφαρμογή είναι ουσιαστική σημασία. Τα κράτη-μέλη λοιπόν και οι δυνατότητε συνεργασία είναι ο σημαντικό παράγοντα. Ένα ερώτημα. Η αξιολόγησή σα για τον ε, προπολογισμό, την συνεισφορά του κοινοτικού προπολογισμού για την ΠΕΣΚΟ. Τα κράτη-μέλη ξέρουμε ότι πολλές φορές έχουν ενδιασμούς για την αποστολή κάποιων αποστολών, αν πρέπει να καταβάλουν το τίμημα τα ίδια. Ένα άλλο ερώτημα είναι αυτό το οποίο αφορά την ε, συνεργασία σε θέματα άμυρας βάσει κοινών πληροφοριών. Με ποιους μηχανισμούς θα ενισχύσετε την διάθεση πληροφοριών από την ΠΕΣΚΟ. Τρίτη ερώτηση. Η ΠΕΣΚΟ θα υποστηρίζει και σχέδια ε, συνεργασία σε τοπικό επίπεδο, φερειπίν, μεταξύ των χωρών της Βαλτικής. Τελικά, αναφέρεται δύο προγράμματα. Την, ε, ε, το κέντρο ενημέρωσης στον κυβερνοχώρο και την γρήγορη ανταπόκριση και αντίδραση σε θέματα που αφορούν τον κυβερνοχώρο. Ε, έχει γίνει λόγος επίσης για τη δημιουργία μιας ε, ε ενότητας που θα ασχολείται με θέματα ετοιμότητας σε στη, για την προσία του κυβερνοχώρου. Αυτό κατά κάποιο τρόπο συνάδει με τα σχέδιά σας. Θα ήθελα να ε, προτείνω, εάν συμφωνείτε, τρεις ερωτήσεις και μετά να απαντήσουν οι προσκεκλημένους. Ο κύριος Πάσκο, ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι υπάρχει ε, μία, ε, κάποια αντίθεση, μια καποια αντιθεση μια διχοτομια που δημιουργείται εδώ. Απ' τη μια έχουμε πει ότι πρέπει να αυξήσουμε τις προσπάθειες σε θέματα ε, ασφάλειας και άμυνας, διότι δεν μπορούμε να επαφιόμεθα πάντα και 100% στους συμμάχους τους Αμερικανούς. Και αν το κάνουμε, θα δημιουργήσουμε και περισσότερους συνδυασμού στου Αμερικανού. Θα πρέπει λοιπόν να το αντιμετωπίσουμε το θέμα αυτό. Από τα σχέδιά σα βλέπω ότι προετοιμαζόμαστε πάλι για διαχείριση κρίσεων. Και διαρωτώ με, πιστεύετε ότι σιγά σιγά η ΠΕΣΚΟ θα μπορούσε να στραφεί μαζί με τον ΝΑΤΟ περισσότερο προς την ε, ε, άμυνα και την πράσινη των συμφερόντων της Ευρώπης, διότι η διαχείριση κρίσεων ίσως δεν είναι κάτι το οποίο είναι τώρα με την κατάσταση της Βαλισσούς τώρα. Βλέπω ότι τα σχέδια και ο τρόπος με τον οποίο έχετε σχεδιάσει τα πράγματα είναι πολύ καλός. Θέλετε πραγματικά να κάνετε συγκεκριμένα πράγματα στα πλαίσια ε, των προβλέψεων σας της ασφάλειας της Ευρώπης, αλλά ε, και πάλι νομίζω ότι είναι πιο ενισχυμένο το σκέλος που αφορά την διαχείριση κρίσεων. Ο κύριος Κάρβερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να φύγουμε ε, από την πολιτική. Έχω τεχνικές ερωτήσεις. Σε ποια φάση βρίσκονται οι σκέψεις για τη συμμετοχή τρίτων χωρών στην ΠΕΣΚΟ. Θα μπορούσατε λίγο αυτό να το αναπτύξετε. Και σε ποιο επίπεδο συνεργασίας περιμένετε να ε, είναι οι χώρες αυτές ε, και χρηματοδοτικά και τεχνικά. Και τρίτον, το ΝΑΤΟ συμμετείχε στη διαδικασία αυτά, αυτή και ποια είναι τα ενεργά μέτρα που λαμβάνονται για να εξασφαλίσουμε ότι δεν υπάρχει επικάλυψη ή σύγκρουση με το ΝΑΤΟ. Έχω άλλους τρεις ακόμα, αλλά είπαμε τρεις-τρεις ερωτήσεις και απαντήσεις μετά, οι υπόλοιποι στη συνέχεια. Αν θέλετε να κάνετε και πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις, έχετε το λόγο αρχίσουμε και πάλι από τον αντιστράτηγο. Ευχαριστώ, σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ για τις ερωτήσεις της. Ο καθένας από εμά θα απαντήσει τις ερωτήσεις που είναι της αρμοδιότητάς τους. το ερώτημα που αφορά τα κράτη-μέλη και τους ενδιασμούς τους να συμμετέχουν σε επιχειρήσεις και αποστολές. Βεβαίως το θέμα είναι και θέμα πολιτικής βούλησης. Αλλά η, η οικονομική υποστήριξη είναι σημαντική και θα πρέπει να πείσουμε τα κράτη-μέλη να συνεισφέρουν. Το ερώτημα είναι διπλό. Έχουμε τον μηχανισμό Ατενά, ο οποίος καλύπτει το κοινό κόστος. Στα πλαίσια της διαδικασίας που έχει συμφωνηθεί και κονδυλίων που, των οποίων η χορήγηση βασίζεται σε κάποια κριτήρια. Ένα άλλο ερώτημα αφορά την αύξηση της αλληλεγγύης όσον αφορά την εφαρμογή. Αυτός ο μηχανισμός προβλέπει συνεισφορά και κονδύλια από τα κράτη-μέλη που χρηματοδοτούν τις αποστολές και τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει όμως και με την αρχή της ελληνικής να καλύψουμε και κάποιε δαπάνε που δεν είχαν καταρχάς προβλεφθεί. Τώρα, για τον εξοπλισμό, για την κατάρτιση των διαφόρων μονάδων προβλεπόντουσαν κάποια κονδύλια, αλλά είναι πολύ υψηλός ο πύχης των προσδοκιών των κρατών μελών και δεν έχουμε υλοποιήσει όλα αυτά τα σχέδια. Φαντάζομαι ότι με την ε, χρηματοδότηση των ε, εκ της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα πλαίσια της ευρωπαϊκής πολιτικής άμεσης και συνεργασίας θα μπορέσουμε να υποστηρίξουμε και τέτοιου είδους επιχειρήσεις και αποστολές ώστε να αμβλύνουμε λίγο το οικονομικό άχθος και τη συνεισφορά την οικονομική των κρατών μελών. Δεύτερο ερώτημα. Για το τι ακριβώς κάνει η ΠΕΣΚΟ, τι είναι. Πρώτα απ' όλα, εργαζόμαστε στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Άμυνας και Συνεργασίας, ασκούμε εξωτερική δράση σύμφωνα με αυτά τα οποία προέβλεπε η συνθήκη και προσπαθούμε να ανταποκριθούμε και σε κάποιες προσδοκίες στον τομέα του στρατιωτικού, αλλά βεβαίως, όπως σας είπα, ασκούμε εξωτερική δράση. Τώρα, η... στα πλαίσια της στρατηγικής μας, ένας από τους τομείς μας είναι η προστασία της Ευρώπης, των πολιτών της Ευρώπης. Σεβόμεθα και αναγνωρίζουμε τον ρόλο του ΝΑΤΟ, συμμαχίας και των κρατών μελών σε θέματα άμυνας. Το λαμβάνουμε αυτό υπόψη, αλλά υπάρχουν στην προστασία της Ευρώπης και άλλα θέματα, θέματα τρομοκρατίας και άλλα θέματα τα οποία δεν είναι ε, δικά μα ή άλλα θέματα τα οποία είναι αποκλειστικά του ΝΑΤΟ. Τώρα εμείς επιλέγουμε να αναπτύξουμε αυτά τα οποία είναι της δικής μας αρμοδιότητας σε εξωτερική δράση. Επιτρέψτε μου ευθύ εξ να υπογραμμίσω το εξή. εάν θα μας οδηγήσει στα αποτελέσματα τα οποία προσδοκούμε η ΠΕΣΚΟ όσον αφορά τη συνεργασία σε θέματα άμυνας και αν θα επιτρέψει ε, στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια της ε, σφαιρικής στρατηγικής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των κρατών μελών. Είπαμε ότι έχουμε μια δεσμευτική συμφωνία εκ μέρους των κρατών μελών και έχουμε διάφορα προγράμματα. Όπως σας είπα, όλα αυτά δεν τα κάνουμε στην ΠΕΣΚΟ ασχολούμενοι μόνο με τα προγράμματα. Τώρα, το θέμα της συνεργασίας σε τοπικό επίπεδο. Εάν δείτε την ΠΕΣΚΟ θα δείτε ότι δεν αποκλείεται διάφορα προγράμματα τα οποία θα υποστηριχθούν να αφορούν ε, συνεργασία σε τοπικό επίπεδο. Αυτό όμως το οποίο στο μέλλον θα κάνει η ΠΕΣΚΟ είναι να έχει ε, σφαιρικά μία πιο συνεκτική προσέγγιση. Δηλαδή, ό,τι έχουμε στην Ευρώπη να είναι πιο ε, διαλειτουργικό, πιο λειτουργικό και πιο γενικό. Αυτό ε, το πρόβλημα θα το λύσουμε αν επικεντρωθούμε μόνο σε περιφερειακή συνεργασία. Τώρα, όσον αφορά τα προγράμματα για τον κυβερνοχώρο και την ασφάλεια. θα πρέπει να καθορίσουμε περαιτέρω και πιο λεπτομεριακά όλα αυτά τα προγράμματα Ξέρουμε ότι ασχολείται με τα θέματα αυτά. Το ΝΑΤΟ ξέρουμε ότι υπάρχει η περίφημη ομάδα ε, που μοιράζεται τέτοιου είδους ε, πληροφορίες. Δεν θα μπορούσα να πω όμως όπως ελέγχθη ότι σχεδόν όλα μας τα προγράμματα αφορούν τη διαχείριση κρίσεων έχουμε και θέματα υποστήριξης προγραμμάτων πυρασφαλείας, θέματα που αφορούν την προστασία γενικότερα και αυτό που κάνουμε και αυτό που θα κάνουμε στο μέλλον θα είναι κάτι το οποίο θα μας ζητήσουν τα κράτη-μέλη. Εμείς βεβαίως παρέχουμε υποστήριξη, αλλά κάποιος πρέπει να μας δείξει τι ακριβώς θέλει. Τώρα, το θέμα του ΝΑΤΟ. Δεδομένου ότι είναι θέμα δημόσια συζήτηση. Εδώ και καιρό. Θα πρέπει να τονίσω τρία πολύ σημαντικά ζητήματα. Πρώτα απ' όλα, fake news και παραπληροφόρηση, δεν μιλάμε για κάτι το οποίο αφορά ε, ανταγωνιστική θέση μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΝΑΤΟ σε τέτοιου είδους θέματα. Διότι στην ε, ε, διακηρύξεις στρατηγικής και της δεκαετίας του 90 και το 2010 γίνεται σαφώς αναφορά στην ε, στρατηγική που πρέπει να αναπτύξουμε για την ευρωπαϊκή ασφάλεια. Και βεβαίως εδώ καλωσορίζουμε τις διατάξεις της ε, ε συνθήκης της Λισαβόνας που μιλά για την ΠΕΣΚΟ και τη δημιουργία της. Δεν βλέπω λοιπόν πού θα πρέπει να υπάρχει αντίφαση ή ανταγωνισμός Λέγεται από κάποιους ότι δεν θα πρέπει στην ΠΕΣΚΟ να γίνεται επικάλυψη του τι γίνεται στο ΝΑΤΟ ή να παρεκκλίνει από την πορεία των πραγμάτων. Θα εξασφαλίσουμε ότι κάτι τέτοιο δεν θα γίνει εάν αναπτύξουμε το σχέδιο ικανοτήτων, αν έχουμε συνεκτική ε, προσέγγιση και αυτό το οποίο γίνεται, αν θέλετε, και στα δύο νόμιμα νομικά πλαίσια θα πρέπει να είναι συνεκτικό. Σε αυτή την περίπτωση δεν θα γίνει ίσως λανθασμένη ιεράρχηση προτεραιοτήτων όπως λέγουν κάτι. Τώρα, τα τρίτα κράτη. Προσπαθούμε να δούμε πώς ε, θα εφαρμόσουμε και σε δεσμικό επίπεδο τις διάφορες ε, διαδικασίες, δηλαδή ποια είναι τα μέλη, τα θεσμικά όργανα τα οποία θα συμμετάσχουν στην όλη διαδικασία. Αυτό είναι κάτι που θα το καθορίσουν τα κράτη-μέλη αργότερα, δεν έχουμε φτάσει ακόμη σε αυτό το επίπεδο. Και όσον αφορά το ΝΑΤΟ, μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι έχουμε σε όλα τα επίπεδα πάρα πολύ ανοιχτό διάλογο στα πλαίσια της κοινή δήλωσης Ευρωπαϊκής Ένωσης ΝΑΤΟ για θέματα που αφορούν την Ευρωπαϊκή Ένωση με το ΝΑΤΟ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία Λέζινγκ, μετά κυρία Γκόμες. Πρώτα κυρία Λέζινγκ, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω γερμανικά. Οπότε βάλτε τα ακουστικά σας. Εντάξει. Η πρώτη μου ερώτηση. Προς τον κύριο Ντομέκ. Δυσκολεύομαι πάντα να κατανοήσω ποιος είναι ο τομέας αρμοδιότητας, ποιες είναι οι αρμοδιότητες δηλαδή της ΠΕΣΚΟ. Δηλαδή θα ήθελα τελικά να καταλάβω ποιος τελικά αποφασίζει για την ετήσια έκθεση στην οποία αναφερθήκατε κι εσείς. Ποιος αποφασίζει για αυτή την έκθεση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας. Ποιος ελέγχει κατά πόσο οι χώρες μέλη τηρούν τα κριτήρια συμμετοχής τους ή όχι. Και αν δεν τα τηρούν, ποιος θα πάει στις χώρες μέλη και θα τους το πει και τι θα κάνει. Δεύτερον, όταν ο οργανισμός διαπιστώνει ότι παραβιάζει τα κριτήρια αυτά μια χώρα, τότε μπορεί να ζητήσει από το Συμβούλιο με ειδική πλειοψηφία να αποκλείσει τη χώρα αυτή από την ε, πολιτική αυτή. Έπειτα, όλα τα στοιχεία προβλέπονται στη συνθήκη της συνεργασίας αυτής ή όχι. Υπάρχουν κάποια που αποκλείονται και αν ναι, ποια είναι αυτά. Και επίσης θέλω να ρωτήσω και κάτι για τα προγράμματα. Αναφερθήκαμε σε, εσείς δηλαδή, αναφερθήκατε σε ομάδες προγραμμάτων, κατηγορίες. Όμως τελικά αυτά τα 17 προγράμματα με αυτά θα ασχοληθούμε ή μπορεί να υπάρξουν και περισσότερα από 17 στο μέλλον και αν ε, ναι, τι προγράμματα θα προσθεθούν σε αυτά τα 17. Τα προγράμματα στα οποία αναφερθήκατε εσείς λοιπόν, θα είναι αυτά τα 17 ή θα υπάρξουν και άλλα. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Η κυρία Γκόμες. Θέλω να επανέλθω λίγο. Θα ήθελα να μιλήσουμε λίγο για αυτή την ενίσχυση της αλληλεγγύης. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει προτείνει πολλές φορές μέχρι τώρα ότι θα υπάρχουν διαφορετικές συνεισφορές. Δηλαδή μια χώρα μπορεί να προσφέρει δυνάμεις, ανθρώπινο δυναμικό δηλαδή, άλλες χώρες μπορεί να προσφέρουν χρήματα, αν δεν είναι έτοιμες να προσφέρουν στρατιώτες. Ίσως αυτός θα είναι ένας καλός τρόπος για να ενισχυθεί η αλληλεγγύη στα πλαίσια της πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Τώρα, η σημασία που έχει ο κυβερνοχώρος. Εντάξει, δεν μπορώ να φανταστώ κανέναν τομέα της ε, ζωής μας και πόσο μάλλον της ασφάλειας και της άμυνας που να μην έχει ως πολύ σημαντική διάσταση τον κυβερνοχώρο. Και γνωρίζουμε βέβαια ότι χώρες μέλη έχουν διαφορετική αντίληψη και διαφορετικά επίπεδα ε, προστασίας ικανοτήτων. Πρέπει όμως να μπορούμε να κάνουμε την ε, διαφορά, όχι μόνο για τις χώρες που συμμετέχουν, αλλά και για άλλες. Η ερώτησή μου πάντως είναι, μπορούμε να βελτιώσουμε, να κάνουμε τη διαφορά, αν συνεχίζουμε να αγνοούμε τους τρόπους με τους οποίους έχουμε αφοπλιστεί. Πώς δηλαδή επιτρέψαμε στους αυτούς μας να κυριαρχηθούμε, να ελεγχθούμε από ξένες εταιρείε που ελέγχουν βασικές υποδομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ενέργεια, για παράδειγμα, χτες αναφέρθηκα σε αυτό. Την παραγωγή και την διανομή της ενέργειας. Στη χώρα μου, στην Πορτογαλία, ιδιωτικοποιήθηκε η ενέργεια από την Τρόικα και τώρα είναι στα χέρια, ο έλεγχος τους δηλαδή, στα χέρια του Κινέζικου Κομμουνιστικού Κόμματος. Έχει γίνει ιδιωτικοποίηση λοιπόν πολλών τέτοιων βασικών ε, υποδομών, ενεργειακών πάρκων στην Ευρώπη από ιδιωτικές εταιρείες, κινέζικες ή άλλες και πολλά λιμάνια. Με τρόπο που όπως εκείνη με την Ερικά Σπαβιλά που από ό,τι φαίνεται επέτρεψε στους Ρώσους να επηρεάσουν τις αμερικανικές ε, εκλογές. Έχουμε μια χαρτογράφηση όλων αυτών. Μπορούμε να μιλάμε σοβαρά για ασφάλεια στον κυβερνοχώρο αν εξακολουθούμε να αγνοούμε αυτή τη διάσταση. Και τέλος, μια που υπάρχει και το Brexit και έχουμε τις επιπτώσεις στα πυρηνικά. Ξέρω ότι είναι κάτι που βγήκε από την Ευρική οι πτώσεις όμως υπάρχουν. είναι αρνητικές. Έτσι και αλλιώς ε, τα πυρηνικά δεν νομίζω ότι ε, βοηθούν τις ευρωπαϊκές χώρες στην άμυνά τους. Πάντως, αυτός ο προβληματισμός έχει μπει καθόλου και συζητιέται καθόλου μεταξύ των στρατιωτικών στην Ευρώπη. Λίτς, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ για τις πληροφορίες που μας δώσατε. Η ΠΕΣΚΟ πιστεύω ότι είναι ένα καλό μέσο για να προχωρήσουμε περισσότερο, να βελτιωθεί η κατάσταση και νομίζω ότι αυτή είναι η επίσημη θέση και η δικιά μου που, είναι, που είμαι Γερμανός σοσιαλιστής αλλά και άλλων Γερμανών είναι κάτι το οποίο θέλαμε εδώ και πολύ καιρό. Αλλά εντάξει, ξέρω ότι η ΠΕΣΚΟ δεν είναι ακριβώς ε, ο ενιαίος ευρωπαϊκός στρατός. Για να επανέλθω στο θέμα του κυβερνοχώρου. Αποτελεί μια τεράστια ευκαιρία για να υπάρξει εναρμόνιση στην Ευρώπη και της στρατιωτικής διάστασης, αλλά για να μπορούμε και μαζί να έχουμε μία δομή στην οποία θα λάβουμε υπόψη μας τις διαφορετικές νοοτροπίες που επικρατούν. Πώς θα λειτουργήσουν διαφορετικοί μηχανισμοί συγχρόνως, όπως θέλουμε να το κάνουμε με το στρατό. Άρα λοιπόν στον τομέα της προστασίας του κυβερνοχώρου μπορούμε να διδαχτούμε πολλά και για την στρατιωτική διάσταση. Τώρα, για να υπάρξει περισσότερη συνένεση στην Ευρώπη, περισσότερη εναρμόνιση, σίγουρα η ΠΕΣΚΟ αποτελεί ένα σημαντικό μηχανισμό, όπως και το Ταμείο που είπατε. Τι μπορεί να κάνει το Κοινοβούλιο, μακροπρόθεσμα δηλαδή, τι απόφαση πιστεύετε ότι είναι εφικτή, αλλά και είναι ανάγκη δικιά μας η Επιτροπή να στηρίξει. Τι μεταρρυθμίσεις πιστεύετε δηλαδή ότι πρέπει να γίνουν στα επόμενα 5-10 χρόνια και θα έπρεπε να προωθήσουμε. Πρόεδρος. Έχω εγγραφεί κι εγώ στον κατάλογο. I mean, um... Και έχω μια πολύ απλή ερώτηση. Βλέπουμε την πολιτική φιλοδοξία βλέπουμε και τη συνθήκη της Λισαβόνας. Από την άλλη όμως βλέπουμε επίσης μεγάλες ανησυχίες από τους εταίρους μας στο ΝΑΤΟ. Αν δούμε την ΠΕΣΚΟ ε, πιο στενά, θεωρώ ότι η κίνησή της έγινε με πολύ βραδείς ρυθμούς. Το χρονοδιάγραμμα λοιπόν ποιο είναι, πότε αναμένεται να πάρει σάρκα και ωστά αυτό που τώρα μάλλον είναι σε επίπεδο προθέσεων. Δεύτερον, ποια είναι τα εμπόδια προς το δρόμο αυτό. Ποια θεωρείτε εσείς αυτή τη στιγμή τα μεγαλύτερα εμπόδια. Και σε ποιο βαθμό πρέπει να ληφθούν αποφάσεις και ποιες είναι αυτές οι αποφάσεις. Μιλήσατε για το μηχανισμό Ατένα Αναφερθήκατε σε διάφορα projects, έργα, αλλά δεν έχει αποφασιστεί ακόμα ο προϋπολογισμός. Ποιο είναι το πρώτο βήμα που πρέπει να ακολουθήσει τώρα για να θεωρήσετε εσείς ότι υπάρχουν τα πρώτα επιτεύγματα και ποιες είναι οι αποφάσεις που πρέπει να ληφθούν έτσι ώστε να ξεκινήσει όλη αυτή η προσπάθεια ουσιαστικά. Αποφασίστε ποιος θα απαντήσει. Ξέρετε πώ σε τα κοινοβούλια κάνουμε γενικέ ερωτήσει και δεν λέμε προ ποιον ομιλητή απευθυνόμαστε. Θέλετε να ξεκινήσετε εσεί ε, στρατηγέ, μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ουσιαστικέ και βαθίε ερωτήσει σα. Ε, αν μου επιτρέπετε, για το μηχανισμό Αθένα, πραγματικά συμφωνώ, δεν ήταν ερώτηση, ήταν δήλωση μάλλον. Υπάρχουν διάφορες διαδικασίες που έχουν τα κράτη-μέλη ε, για να διευρύνουν ε, το μηχανισμό αυτό Αθήνα και το πεδίο εφαρμογή. Και τα κράτη-μέλη συμμετέχουν εθελοντικά, ε, πολύ ελδοφόρα μηνύματα. Αν κάποιος δεν θέλει να συμμετέχει ουσιαστικά επιχειρησιακά, δηλαδή με ένοπλες δυνάμεις, μπορεί να συμμετέχει με άλλες ικανότητες, με υλικό ή με χρηματοδότηση ή με άλλους όρους. Για το θέμα τώρα του μηχανισμού Αθήνα, και πώς ε, βελτιώνεται η αλληλεγγύη και οι μηχανισμοί. Αυτό είναι περίπλοκο. Φυσικά εδώ μιλάμε για κρατικούς πόρους, γιατί χρήματα των κρατών μελών. Δεν είναι από τον κοινό ευρωπαϊκό κορβανά και τα κράτη-μέλη κοιτάνε πάρα πολύ προσεκτικά πώς δαπανώνται αυτοί οι πόροι. Υπάρχουν κάποια κριτήρια για να είναι επιλέξιμα για τη χρηματοδότηση από το μηχανισμό Αθηνά. Και υπάρχει μεγάλη πολιτική βούληση για να διευρυνθεί ε, αυτός ο μηχανισμός χρηματοδότησης ε, ε, για τους περίφημους μάχημους σχηματισμούς. Αυτό δεν χρησιμοποιείται ως εργαλείο. Συνεχίζεται η συζήτηση κατά πόσο το κόστος ανάπτυξης ή και εκπαίδευσης μπορεί να καλυφθεί από εκεί. Στο χρηματοδοτικό μηχανισμό Αθηνά. Και αν πάνε όλα καλά, μπορεί να πείσουμε και τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν ε, αυτή τη δυνατότητα για τη χρηματοδότηση των μάχημων σχηματισμό. Αυτό είναι πολιτική απόφαση. Υπάρχει όμως ένα πρακτικό ζήτημα που αντιμετωπίζω εγώ στη γραμματεία μου ε, και στην επιχειρησιακή διοίκηση για τους μηχανισμούς και τις αποστολές τις εκπαιδευτικές όλο και περισσότερο υπάρχουν ανάγκες εκεί χρηματοδότησης και πολύ τεκμηριωμένες και εμπεριστατωμένες για το υγειονομικό, ας πούμε, για την προστασία των ενόπλων δυνάμεων. Και τα κράτη-μέλη δεν είναι πάντα πάρα πολύ πρόθυμα να βοηθήσουν από τις ίδιες τους τις ικανότητες. Εξού και ε, ανατρέχουμε στο Αθηνά και ε, αναθέτουμε σε εξωτερικούς ορισμένες ικανότητες. Γιατί μπορεί να έχουμε την ικανότητα αυτή, αλλά δεν είναι τόσο φτηνή, είναι ακόμα πιο ακριβή και δεν είναι και τόσο ικανή αυτή η ικανότητα εντό εισαγωγικών, όσο αν την έδιναν τα κράτη-μέλη. Υπάρχει λοιπόν χώρος για βελτίωση ακόμα εκεί, αλλά όπως σας είπα, προσπαθούν τα κράτη-μέλη να δουν πώς μπορεί να αυξηθεί η ευελιξία και να χρησιμοποιηθεί καλύτερα αυτός ο μηχανισμός χρηματοδότησης. Υπάρχουν κάποιες γκρίζες ζώνες που δεν έχουν ακόμα διευκρινιστεί, για να το πω έτσι, απολύτως και πλήρως. Παραμένει κάποια ασάφεια. Το θέμα του Brexit τώρα. Εγώ θα το έβλεπα διαφορετικά τι σημαίνει το Brexit για τις ικανότητες και τη στρατιωτική διάσταση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βεβαίως έχει και περιχυσιακές επιπτώσεις ή μπορεί να έχει, γιατί στο Λονδίνο είναι το επιτελείο που χειρίζεται την κοινή επιχείρηση Αταλάντα. Και επίσης θα πρέπει να αντικατασταθεί κάποια συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου. Το δεύτερο γενικότερο θέμα για τις ικανότητες αν δούμε τον κατάλογο ικανοτήτων για να δηλώσουν τα κράτη-μέλη, τι χρειαζόμαστε για να υποστηρίξουμε ε, τις ε, αποστολές μας, τις ε, στρατηγικές ικανότητες, είναι μεγάλο το μερίδιο του Ηνωμένου Βασιλείου και αν χαθεί αυτό θα υπάρχει έλλειμμα και θα πρέπει να καλυφθεί. Και μετά υπάρχει και το θέμα του προσωπικού των υπαλλήλων. Ε, εγώ έχω 15 ε, αξιωματικούς που εργάζονται στο επιτελείο μου, Βρετανούς και πραγματικά, βέβαια δεν είναι το δικό μου το προσωπικό, αλλά είναι και το στοιχείο αυτό του ανθρώπινου δυναμικού. Η ε, πυρηνική αποτροπή αυτού συνδέεται μάλλον με το πολιτικό σκέλος της επιχείρησης και της άσκησης. Είναι πυρηνικές δυνάμεις στο Ηνωμένο Βασίλειο και η Γαλλία, είναι και μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας μόνιμα μέλη ε, του ΟΗΕ. Άρα είναι πολιτικό μάλλον το θέμα. Σταματώ εδώ και θα δώσω το λόγο στον Χόρχε. Ευχαριστώ. Καταρχάς, όταν λέτε ότι είναι δύσκολο να κατανοήσουμε την ΠΕΣΚΟ, είναι πολλοί οι πολίτες τους οποίους θα πρέπει να το εξηγήσουμε πραγματικά ε, περί τίνος ακριβώς ε, πρόκειται, δεν είστε μόνο εσείς. Ε, υπάρχει εκτίμηση ε, ότι, ε, και την κάνουμε αυτή η αξιολόγηση στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας, και αυτό το τσεκάρουμε ε, ως προς τις 20 δεσμεύσεις των κρατών μελών. Τι έχουν κάνει σε εθνικό επίπεδο, ε, τα δικά τους σχέδια και πώς τα εφαρμόζουν με χρονοδιαγράμματα. Έτσι ώστε να υλοποιήσουν αυτούς τους στόχους. Είναι βάση των πληροφοριών που έχουμε και τις ε, δεσμεύσεις που έχουν συμφωνήσει και αναλάβει οι χώρες μέλη. Είναι ξεκάθαρη λοιπόν αξιολόγηση αυτή. Ε, εμείς κάνουμε την αξιολόγηση ο Οργανισμός Άμυνας, θα τη δώσουμε στην ύπατη εκπρόσωπο, η οποία θα την εντάξει στη δική της αξιολόγηση που εξετάζει άλλα στοιχεία επιχειρησιακά, από την Υπηρεσία εξωτερική δράση και το στρατιωτικό επιτελείο τη Ευρωπαϊκή Ένωση. και αυτά θα τα υποβάλει συνέχεια η κυρία Μογερίνη στο Συμβούλιο. Προηγουμένω, η Στρατιωτική Επιτροπή τη Ευρωπαϊκή Ένωση θα νομοδοτήσει ε, για τις αξιολογήσεις αυτές και με τη σειρά του το Συμβούλιο θα πάρει αποφάσεις συμπεριλαμβανομένης και της απόφαση τι θα την κάνουν την έκθεση αυτή. Αυτό αφορά άμεσα τα κράτη-μέλη και προς εκείνους απευθύνεται. Εγώ δεν θα ανέμενα. Μάλλον η έκθεση κανονικά θα πρέπει να επισημαίνει τα στρεβλά, ε, πού δεν πηγαίνουμε καλά και πού ε, θα προχωρήσουμε καλύτερα για να υλοποιήσουμε τους στόχους που εμείς έχουμε αναλάβει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα από τα προβλήματα για τα κράτη-μέλη θα ήταν ακριβώς αυτό, να, να ποια είναι τα προβλήματα και τα, οι αδυναμίες για να μπορέσουν να τα αντιμετωπίσουν ποια θα είναι στην ΠΕΣΚΟ και ποια γενικότερα στην ΕΠΑ. Εξαρτάται από το επίπεδο της φιλοδοξίας. Αφού συμμετέχουν 25 κράτη-μέλη εκεί από τα 28, ήδη στην ΠΕΣΚΟ, και ένα κράτος μέλος αποχωρεί του χρόνου, Υπάρχει ένα που έχει προχωρήσει σε opt-out, εξαίρεση, από την ΕΠΑ. Άρα, στο μέλλον, στο πλαίσιο ΠΕΣΚΟ, θα έχουμε πάρα πολύ μεγάλη συνεργασία ε, για την ΕΠΑ. Ποια είναι τα σημερινά έργα που υπάρχουν 17 τον αριθμό και πρόκειται στην απόφαση του Συμβουλίου την άλλη εβδομάδα αυτά να, να συγκεκριμενοποιηθούν και να επισημοποιηθούν. Θα υπάρξουν και περισσότερα. Ναι, τα κράτη-μέλη έχουν ζητήσει να υπάρξει ένα δεύτερο κύμα, όπως το είπαμε, κατά τη διάρκεια του έτους ποια είναι αυτά που θα προσθεθούν. Και πάλι αυτό είναι ε, απόφαση στα χέρια των κρατών μελών. Εμείς μαζί με τη γραμματεία της ΠΕΣΚΟ ε, έχουμε ως αποστολή να δούμε αν ανταποκρίνονται αυτά τις προτεραιότητες της ΕΠΑ και αν λαμβάνονται υπόψη και άλλα στοιχεία. Μπορούν να υποφεληθούν από το Ευρωπαϊκό Ταμείο αν χρειάζεται χρηματοδότηση. Γίνεται έρευνα για τη βιομηχανική ανάπτυξη. Τι γίνεται με, την ε, ανάπτυξη των ικανοτήτων και πώς εγγράφονται στο γενικότερο πλαίσιο. Στο μέλλον, θα έχουμε μια συντονισμένη ετήσια αναθεώρηση και επιθεώρηση ε, της άμυνας και θα λέμε εδώ υπάρχουν αδυναμίες, εδώ υπάρχουν προβλήματα, κατακαιρματισμοί, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συντονιστούν περισσότερο για να έχουμε στο μέλλον καλύτερο αποτέλεσμα στο τέλος. Για το σχέδιο ανάπτυξης ικανοτήτων και τη σημασία του κυβερνοχώρου. Αυτό που με ρωτάτε τι είναι. Τι μπορούμε να κάνουμε για να βελτιώσουμε τον έλεγχο των εθνικών δυνατοτήτων. Όπως ξέρετε, τα κράτη-μέλη δεν θέλουν να ελέγχονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ούτε να παρακολουθούνται για το πώς χρησιμοποιούν τους εθνικούς τους πόρους. Είναι αμυγός εθνικό αυτό το ζήτημα. Και αυτό είναι πολύ εκτός του δικού μας ε, πεδίου δραστηριοτήτων και των εξουσιών μας και αρμοδιοτήτων μας. Εγώ σε δύο τομείς μπορώ να προσφέρω. Στην ε, κατάρτιση και εκπαίδευση και στις ασκήσεις. Και εκεί ε, τα καλά νέα είναι ότι την περασμένη εβδομάδα αποφασίσαμε βάσει μιας μελέτης που αναθέσαμε με, βοήθεια από τη Στρατιωτική Επιτροπή να έχουμε στη σχολή Εθνικής Αμήνης στην Ευρωπαϊκή ε, ε, Εκπαίδευση για την ΕΠΑ και οι ασκήσεις. Έτσι ώστε να μπορούμε να πιστοποιούμε ε, τις δεξιότητες και τις ικανότητες του προσωπικού παντού στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να μην χρειάζεται να γίνεται αυτό ξεχωριστά σε κάθε χώρα μέλος. Και από την άλλη υπάρχει μια ανάγκη κοινή προσπάθειας στην έρευνα. Στην κοινή έρευνα ακριβώς στον κυβερνοχώρο που είναι κρίσιμος τομέας οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων μας το ανέθεσαν αυτό από το 2013, αλλά και πάλι ο κυβεροχώρος είναι πάρα πολύ ευαίσθητος τομέας, γιατί σας αναγκάζει να ε, δείχνετε τις ευάλωτες πτυχές σας και τις τροτές. Ε, αλλά αυτό θα πρέπει να το δούμε. Κύριε Λίτς, απαντώντας και σε εσάς, ο κυβερνοχώρο είναι πραγματικά ένας τομέας που μπορούμε να το ε, εναρμονίσουμε όλο αυτό. Τι θα μπορούσατε να έχετε κάνει εσείς. Όπως σας είπα, η ΣΕΝΤΕ ήταν πολύ ε, κρίσιμη, όχι μόνο για την ΠΕΣΚΟ, υπό Επιτροπή σας, αλλά για όλες τις προτάσεις. Γιατί σε κάποιο βαθμό η ΠΕΣΚΟ είναι ε, η άλλη όψη του Οργανισμού Άμυνα στη Συνθήκη. Από σας παρακαλώ πραγματικά να παρακολουθείτε ε, τις εξελίξεις. Έρχομαι τώρα στην ερώτηση του κυρίου Έλερ για την βραδία εκκίνηση των διαδικασιών της ε, συνεργασίας ΠΕΣΚΟ και εδώ θα κλείσω από εκεί που ξεκίνησα. Το σημαντικό εδώ δεν είναι τα project, τα έργα. Αυτό που πρέπει να επιτύχουμε είναι το εξής. Τα κράτη-μέλη πραγματικά να αρχίσουν να σχεδιάζουν από κοινού. Και τα αμυντικά τους σχέδια δεν καταρτίζονται εν μία νυχτή. Βρισκόμαστε στην αρχή και μόνο μιας μακράς διαδικασίας και μιας μακράς εργασίας για όλη την Ευρώπη. Και σιγά σιγά τι θα πρέπει να δούμε τα επενδυτικά του σχέδια, τα σχέδια για την ανάπτυξη ικανοτήτων, τους στόχους να μπορούν να στέλνουν και να αναπτύσσουν δυνάμεις ε, σε αποστολές, να μην τα βλέπουν αυτά αμυγός εθνικά. Η Πέσχο δηλαδή, τι σημαίνει να πρέπει να εγκαταλείψουμε την ιδέα ότι η άμυνα είναι κάτι αμυγός εθνικό και να πάμε σε μια πιο ολοκληρωμένη προσέγγιση πανευρωπαϊκή. Και όσο προχωρούμε θα φτάσουμε εκεί, αλλά το σημαντικότερο είναι αν αρχίζουμε από κοινού να επενδύουμε, να σχεδιάζουμε, να αναπτύσσουμε τα έργα και αυτό θα είναι το αποτέλεσμα. Το ξέρω ότι μας αρέσουν οι γρήγορες επιτυχίες και να αποδώσει κάτι γρήγορα, αλλά αυτό μας ενδιαφέρει είναι σιγά σιγά να αποφύγουμε τον κατακαιρματισμό και να ε, συνεισφέρουν τα κράτη προς την διακατεύθυνση. Ε, αν το κάνουμε αυτό πραγματικά θα είναι ένα βήμα πρόοδου. Να τελειώσει ο στρατηγός. Ναι, θα ήθελα λίγο να συμπληρώσω αυτό που είπε ο Χόρχε. Για πολλά χρόνια έκανα αμυντικό σχεδιασμό στην πρωτεύουσα της χώρας μου και ξέρω πόσο περίπλοκο είναι να βρούμε κοινό έδαφος για μια κοινή ανάπτυξη γιατί οι κύκλοι προγραμματισμού της κάθε χώρας διαφέρουν από την διπλανή. Αυτός ο συντονισμένος τρόπος ετήσιας αναθεώρησης θα βοηθήσει τα κράτη-μέλη να συμπλησιάσουν ε, το δυναμικό τους για ε, τις προμήθειες και τα σχέδιά τους αν είναι πλήρως διαφανή. Αυτά ε, είναι πιο μακροπρόθεσμα για το κοινοβούλιο και το ρόλο του. Πώς να το πω. Εγώ δεν τα ξέρω από μέσα πώς λειτουργεί το κοινοβούλιο και η υποεπιτροπή σας, αλλά ένα σημαντικό ζήτημα για τις συζητήσεις είναι οι χρηματοδοτικοί μηχανισμοί και Ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει, έχει γι' αυτό και το Κοινοβούλιο έχει ρόλο να διαδραματίσει. Κάτι άλλο όμως που με απασχολεί πολύ και το βλέπω όταν πηγαίνω να επισκέπτομαι ε, τα διάφορα κράτη-μέλη της Ένωσης και συναντώ πολίτε, είναι ότι ο κόσμος δεν γνωρίζει τι γίνεται εδώ, τι κάνουμε. Εσείς είστε πολιτικοί, εσείς είστε βουλευτές και όσα περισσότερα γνωρίζετε, τόσο καλύτερα μπορείτε να ενημερώνετε τον κόσμο οι ίδιοι για το ευρωπαϊκό αμυντικό εγχείρημα, το τι είναι και κυρίως τι δεν είναι. Και αυτό το θέμα τα επόμενα έτη θα είναι ακόμα πιο σημαντικό από τα υπόλοιπα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε πολύ για τα συμπεράσματά σας. Ε, μικρά βήματα μας κάνουν να προχωρούμε. Άλλες ερωτήσεις. Όχι εντάξει, τότε θα διακόψουμε για λίγο. Η κυρία Φωτίγκα ήρθε και θα αρχίσουμε πάλι στις 11.30 όπου θα έχουμε τον Αντιπρόεδρο της Ουκρανίας. Μην ε, φύγετε. Colleagues, please be seated. Αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε παρακαλώ. Καθίστε παρακαλώ αγαπητοί συνάδελφοι. Ευχαριστώ. Περνάμε στο επόμενο σημείο της ημερήσιας διάταξης που είναι το τελευταίο ουσίας αυτή της δίμερης συνεδρίασης της Υποπιτροπής μας Ασφάλειας και Άμυνας. Το θέμα μας είναι η εξελισσόμενη κατάσταση ασφάλειας στην Ανατολική Ουκρανία και ποιες είναι οι προοπτικές για την αποστολή την ειρηνευτική του ΟΙΕ στην περιοχή. Χαίρομαι πάρα πολύ λοιπόν που έχω το προνόμιο να υποδεχτώ εδώ την κυρία Ιβάνα Κλίμπους Τζιντζάτσε που είναι η αντιπρόεδρος της κυβέρνησης της Ουκρανίας υπεύθυνη για την ευρωατλαντική ολοκλήρωση. Συνοδεύεται από τον γνωστό σε μας πρέσβη της Ουκρανίας, τον κύριο Μεκατοτσίτσκι. Χωρίς άλλη καθυστέρηση λοιπόν, ξέρω ότι ο χρόνος σας είναι πολύτιμος, οπότε είσαστε και ο πιο κατάλληλος άνθρωπος για να μας μιλήσει για αυτά τα θέματα που μας ενδιαφέρουν. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι ευγνώμων για την ευκαιρία αυτή που μου δίνετε και για την πρόσκλησή σας να έρθω και να απευθυνθώ εδώ στους ευρωβουλευτές της Υποπιτροπής σας για την ασφάλεια και άμυνα. Υπενθυμίζω ότι είχα την τιμή να έρθω εδώ και πριν ακριβώς από ένα χρόνο. Τότε που είχαμε ξαφνική επιδείνωση της κατάστασης στην Ανατολική Ουκρανία το τέλη του Φεβρουαρίου του 2017. Θα αρχίσω από το ότι εμείς οι Ουκρανοί στην Ουκρανία καταλαβαίνουμε πάρα πολύ καλά ότι η δημοκρατία είναι κάτι για το οποίο πρέπει να αγωνιστεί κανείς και πρέπει να προστατεύει. Και αυτό το μάθαμε με την σκληρή εμπειρία που έχουμε τα τελευταία χρόνια μετά από την επίθεση της Ρωσικής Ομοσπονδίας που προσάρτησε την Ανατολική Ουκρανία και στη συνέχεια επιτέθηκε και σε, την Κρυμαία και στη συνέχεια επιτέθηκε στα ανατολικά τμήματα της χώρας, της Ουκρανίας. Το καταλαβαίνουμε λοιπόν αυτό και αντιλαμβανόμαστε απόλυτα την ανάγκη αυτή προστασίας της δημοκρατίας. Το σπαζόμαστε. Τώρα, εμείς ακριβώς με τόσα έχουμε κάνει, ακριβώς ε, αυτό δείχνουμε ότι σπαζόμαστε αυτή την ιδέα. Όμως, τα χαρακτηριστικά ε, από τότε που ανακτήσαμε την ανεξαρτησία μας ήταν παρέμβαση και ε, Δίστηση σε διάφορα επίπεδα της Ρωσικής ομοσπονδίας ακόμα και στην ε, θεσμική οικοδόμηση της χώρας. Προσπάθησαν να επιβληθούν. Γι' αυτό λοιπόν και εμείς καταλαβαίνουμε και πάλι από την εμπειρία μας ότι η Ρωσία προσπαθεί να ελέγξει τελικά και πάλι τη χώρα. Ισχύει αυτό για την Ουκρανία, το καταλαβαίνουμε. Στόχος μας, ο στόχος τους μάλλον δεν είναι μόνο η Ουκρανία. Δυστυχώς οι ορέξεις του Κρεμλίνου είναι πολύ μεγαλύτερες και επεκτείνονται σε ολόκληρο το δυτικό κόσμο, σε ολόκληρη αυτή την ενότητα δυτικών χωρών και έτσι επιδεινώνεται η κατάσταση με τις παρεμβάσεις αυτές της ε, Ρωσίας κατά του διεθνούς δικαίου. Και είναι κάτι λοιπόν που συμβαίνει όχι μόνο στην Ουκρανία, αλλά σε ολόκληρο τον κόσμο. Το τελευταίο καιρό εξακολουθούμε να μετράμε τις απώλειές μας και εξακολουθούμε να βλέπουμε τους στρατιώτες μας να πεθαίνουν στο μέτωπο, στην γραμμή δηλαδή που ελέγχεται και κατέχεται στα ανατολικά της Ουκρανίας από τη Ρωσία. Ήδη χάσαμε 22 στρατιώτες τώρα το 2018 και είχαμε και 97 τραυματισμένους. Λοιπόν, όλες αυτές οι διαπραγματεύσει που έχουν γίνει για κατάπαυση πυρό παραβιάζονται, συνεχώς παραβιάζονται από τους ε, όσους ελέγχει η Ρωσική Ομοσπονδία τους μισθοφόρους της Ρωσικής Ομοσπονδίας. Βέβαια, οι μάχες ε, καταλήγουν στο να βλέπουμε καταστραμμένες υποδομές, σπίτια, δρόμους και από εκτίμηση του Υπουργείου μας Άμυνας βλέπουμε ότι έχουμε καταστροφές 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων στο ανατολικό τμήμα της χώρας. Και όλα αυτά συνοδεύονται και με έναν πόλεμο πληροφόρησης. Τα ξέρετε κι εσείς από τις χώρες σας τι σημαίνει αυτό από πλευράς της Ρωσίας και της ρωσικής προπαγάνδας η οποία διαχέεται όχι μόνο στα μέσα ενημέρωσης αλλά και σε διάφορα think tanks, στο facebook, σε διαδικτυακές ε, σελίδες κλπ. Υπάρχει λοιπόν ε, παραπληροφόρηση η οποία έχει στόχο να μας απομονώσει από τη διεθνή κοινότητα και από τους συμμάχους μας, με τους οποίους είμαστε ενωμένοι όσον αφορά την επίθεση αυτή της Ρωσίας ε, στο διεθνές δίκαιο. Ξέρουμε ότι αυτό είναι ένα μέσο που χρησιμοποιούν και προσπαθούν έτσι να κατακτήσουν ολόκληρο το κόσμο. Δεν περιορίζονται στην Ουκρανία. Αξιότιμοι ευρωβουλευτέ, μέλη της Επιτροπής ΕΔΕ. Η κατάσταση όσον αφορά την ασφάλεια στα κατεχόμενα της Ουκρανίας παραμένει πάρα πολύ ρευστή. Και δεν βλέπουμε καμία επιθυμία ούτε δέσμευση από την Ρωσική Ομοσπονδία να τηρήσει τις συμφωνίες του Μίνσκ. Αντίθετα, οι δράσεις τους είναι εκτός πλαισίου συμφωνίας του Μίνσκ. Και δεν μένουν στα θέματα τα οποία συζητήθηκαν στο Μίνσκ και συμφωνήθηκαν προκειμένου να υπάρχει διάλογος. Δεν υπάρχει επίσης κατάπαυση πυρός ...που να τηρείται. Εξακολουθεί η Ρωσία να ε, παρεμβαίνει και να επιτίθεται και δεν ε, επιτρέπει ούτε καν το 7 ημέρο εκείνο κατάπαυσης ε, πυρός που είχαμε συμφωνήσει. Δεν υπάρχουν καν και δραστηριότητες ε, καταστροφής των ε, ναρκών που είχε συμφωνηθεί με την ε, Ρωσία, που σημαίνει ότι είμαστε η χώρα στον κόσμο της περισσότερες νάρκες. Σήμερα λοιπόν αρχίζουμε να προσπαθούμε την καταστροφή των ναρκών σε όλες αυτές τις περιοχές που είχαν μπει οι νάρκες κοντά στην γραμμή των κατεχομένων. Δεν έχουμε καν ε, την ε, πρόσβαση της αρμόδιας υπηρεσίας ε, του ΕΕ, ούτε καν, όχι μόνο στα κατεχόμενο, αλλά ούτε καν και στην γραμμή διαχωρισμού. Αποσύρθηκε και από το κοινό κέντρο ελέγχου και συντονισμού η Ρωσία το Δεκέμβριο, κάτι το οποίο υπονομεύει το έργο της αποστολής εποπτείας. Με σκοπό η Ουκρανία να έχει διάλογο με την Ρωσία υπό ρωσική ηγεσία. και να φανεί ότι η εμπλοκή της Ρωσίας είναι πολύ μικρότερη από αυτή που πραγματικά είναι. Για τους Ουκρανούς καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι και πολύ συναισθηματικά φορτισμένα. 75 από τους ομήρους μας επέστρεψαν, αλλά δυστυχώς μετά από αυτό δεν απελευθερώθηκαν άλλοι όμοιροι και ακόμα και αν βλέπουμε κάποια δείγματα αισιόδοξα, δεν έχει υπάρξει αλλαγή, ούτε και όσον αφορά τους αγνούμενους, Με πρόσβαση ανθρωπιστικών οργανώσεων στα κατεχόμενα. Έχουμε και δυσκολίες με την εφαρμογή προγραμμάτων όσον αφορά την προμήθεια νερού και ηλεκτρισμού. Διακόπτη η Πρόεδρος. Μπορείτε να μιλάτε λίγο πιο αργά για να σας προλαβαίνουν και οι διερμηνείς, λέει η Πρόεδρος. Οι υποδομές στα κατεχόμενα, όπως είπα, έχουν καταστραφεί σημαντικά. Το 2017 θα σας δώσω κάποια νούμερα τώρα. 535 σπίτια και υποδομές καταστράφηκαν 98 ε, μη στρατιωτικοί σκοτώθηκαν και 552 τραυματίστηκαν στα κατεχόμενα. Η Ρωσία συνεχίζει να καταστρέφει και το βιομηχανικό δυναμικό του Ντονμπάς με ρήπανση και με καταστροφή των ε, πιο πολύτιμων βιομηχανικών υποδομών εκεί. Το 1 τρίτο του δυναμικού του βιομηχανικού στον Τονμπάς έχει καταστραφεί και μεταφερθεί στη Ρωσική Ομοσπονδία. Και είναι μια από τις πιο σημαντικές βιομηχανικές μονάδες που είχαμε στη χώρα. 67% των βιομηχανικών δυνατοτήτων της περιοχής του Ντονιέσκ. Είναι στα κατεχόμενα και το 1 τρίτο σας είπα έχει ήδη μεταφερθεί στη Ρωσική Ομοσπονδία. Και υπάρχουν και μεγάλες καταστροφές επιτόπου. Δεν υπάρχει λοιπόν πρόοδος ούτε και για το θέμα των τοπικών εκλογών στον Τονμπάς. τη στιγμή που μονομερός η Ρωσία αποφασίζει να αναγνωρίσει τις ταυτότητες που εκδίδουν παράνομες αρχές στα καταχώμενα. Το ρίζιμιές και οι απώλειες του πολέμου αυτού που είναι στη χώρα μας είναι πάνω από 16.000 άνθρωποι που έχουν χάσει τη ζωή τους και 3.753 έχασαν ε, τη ζωή τους πολεμώντας. Και πάρα πολύ τραυματίστηκαν όλο αυτό το διάστημα. Η πρόκληση αυτή της Μόσχας ανάκασε την Ουκρανία να προσαρμοστεί ανάλογα με την κατάσταση επιτόπου και γι' αυτό και πρόσφατα το κοινοβούλιο μας ψήφισε ένα νόμο για την επανένταξη που υπεγράφηκε από τον πρόεδρο της Ουκρανίας που θεωρεί τη Ρωσία επιθετική δύναμη. Και αυτό βάσει της κατάστασης που έχουμε σήμερα στο Τανμπάς, που παραβιάζει κατάφορα το διεθνές δίκαιο. Ο νόμος αυτός όμως δεν σημαίνει ότι εμείς δεν θέλουμε να τηρήσουμε τις συμφωνίες του Μίνσκ. Και προσπαθούμε να υιοθετήσουμε ρυθμίσεις για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κόσμου στα κατεχόμενα και να ρυθμίσουμε το νομικό καθεστώς των κατεχομένων. Όλες αυτές οι δράσεις και η κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε στα ανατολικά της Ουκρανίας μας αναγκάζει να αρχίσουμε και πάλι τις συζητήσεις για την ανάπτυξη ειρηνευτικής δύναμης στα εδάφη της Ουκρανίας. Θέλω να επενθυμίσω και να υπογραμμίσω ότι ήταν η Ουκρανική Προεδρία, ο Πετροσέγκο, όπου την άνοιξε το 2015 έστειλε έτοιμα στο Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ και το Πρόεδρο του Συμβουλίου Ασφαλείας για την ανάπτυξη ειρηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ στα κατεχόμενα εδάφη του Ντονμπάς. Και πάντα υποστηρίζαμε μια σαφή θέση για ειρηνευτική αποστολή και την ανάπτυξή της στα ουκρανικά εδάφη. Πρέπει να αναπτυχθεί με την συμφωνία και αποκλειστικές διαβουλεύσεις με την Ουκρανική πλευρά. Πρέπει να αποσυρθούν όλες οι κατεχόμενες δυνάμεις και οι μισθοφόροι και τα όπλα από τα δάφη της Ουκρανίας και πρέπει να υπάρξει αποτελεσματικός έλεγχος των συνόρων Ουκρανίας ε, ε, Ρωσίας, 490.000 χιλιόμετρα. Μιλάμε για αποστολές που έρχονται στην Ουκρανία. Άλλες 74 τέτοιε αποστολές πέρασαν από το κομμάτι που δεν είναι ελεγχόμενο, φέρνοντας ε, όπλα, εξοπλισμό, μισθοφόρους. Έτσι ακριβώς είναι που η Ρωσία διασφαλίζει τη στρατιωτική της παρουσία επιτόπου στα κατεχόμενα της Ουκρανίας. Η απόφαση υπέρ της παρουσίας ειρηνευτικής δύναμης πρέπει να συμπεριλάβει και την έννοια ότι δεν πρέπει να συμμετέχουν σε αυτή ε, εκπρόσωποι προερχόμενοι από την πλευρά που έχει επιτεθεί στην Ουκρανία. Συνεπώς, είναι σημαντικό για μας να εισακουστούμε από τους εταίρους μας και να έχουμε κοινή θέση όσον αφορά τον τρόπο και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιήσει ο ΙΕ, τι εργαλεία θα χρησιμοποιήσει προκειμένου να καταλήξουμε στην ανάπτυξη ειρηνευτικής δύναμης εκεί αγαπητοί ευρωβουλευτές μέλη του, της Επιτροπής ΣΕΝΤΕ, δεν μπορώ να δεχτώ την κατάσταση αυτή της παράνομης προσάρτησης της Κρυμαίας. Τα τελευταία χρόνια η παρουσία της Ρωσίας στην Χερσόνησο έχει σαν αποτέλεσμα να κάνει την τουριστική αυτή περιοχή μια βαριά εξοπλισμένη στρατιωτική βάση. Επιδεινώνεται η κατάσταση και όσον αφορά την ασφάλεια και όσον αφορά την ε, προστασία ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Το καθεστώς το οποίο κυβερνάει την παράνομα ε, προσαρτημένη Κρυμαία πιέζει ψυχολογικά με κρατήσεις, ε, με βασανισμούς είναι πολιτική της Ρωσικής Ομοσπονδίας αυτή. Θα θυμόσαστε ότι οι Ταρτάροι, που είναι αυτόχθονος πληθυσμός στην ε, Κρυμαία, θεωρήθηκαν από το 2016 παράνομοι. Το κοινοβουλίο τους, δηλαδή η Βουλή που είχαν οι Τάρταροι εκεί. Υπάρχουν λοιπόν διωγμοί τους θεώρησαν εξτρεμιστές. Μετά την προσάρτηση της Κρυμαίας επίσης, η Ρωσία ξεκίνησε να προσπαθεί να αφαιρέσει κάθε στοιχείο ουκρανικότητα στην περιοχή. Η Ρωσική Ομοσπονδία επίσης φέτος έχει εγκρίνει 2.000 διαφορετικές ρυθμίσεις προσπαθώντας να ενσωματώσει την Κρυμαία στο νομοθετικό της πεδίο και με 15 συνταγματικούς νόμους που ενέκρινε η Ντούμα. Έτσι παραβιάζει 407 διαφορετικές συνθήκες η Ουκρανία θα συνεχίσει να προσφεύγει στα διεθνή δικαστήρια κατά της Ρωσίας, η οποία παρεβιάζει διάφορες διεθνείς συμβάσεις και ελπίζουμε όντως να προσταχθεί στη δικαιοσύνη η Ρωσία. Θέλω να επαναλάβω ότι η Ρωσία αποτελεί απειλή όχι μόνο για την Ουκρανία, όχι μόνο για τη Γεωργία ή τη Βολδαβία αποτελεί απειλή και για τις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τις χώρες που ασπάζονται τις δυτικές αρχές. Δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ο Πούτιν προέρχεται από την Κακεμπέ και εξακολουθεί να είναι άνθρωπος Κακεμπέ. Ο τρόπος που συμπεριφέρονται αυτοί οι άνθρωποι είναι ότι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν τις αδυναμίες των άλλων και εκμεταλλεύονται αυτές τις αδυναμίες, τους ελέγχουν και ακριβώς αυτό είναι που κάνει η ρωσική πολιτική απέναντι σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες. Η χρηματοδότηση διαφόρων πολιτικών κομμάτων, για παράδειγμα, είτε είναι της δεξιάς είτε είναι της αριστεράς στην Ευρώπη, από την ε, Ρωσία, ε, προσπαθούν να σφετεριστούν ολόκληρα κόμματα, παραστρατιωτικές ομάδες. Προσπαθούν με προπαγάνδα, με τα μέσα ενημέρωσης, να φτάσουν σε διάφορες κοινότητες, κοινωνίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και να τις επηρεάσουν. Με αυτόν τον τρόπο η Ρωσία επιτίθεται στην διεθνή κοινότητα σήμερα. Εμείς λοιπόν Ελπίζουμε ότι θα παραμείνουμε ενωμένοι η Ευρωπαϊκή Ένωση διατλαντικά με τον Καναδά, τις Ηνωμένε Πολιτείε, ότι όλοι ενωμένοι θα διασφαλίσουμε η Ρωσία να μην μπορέσει να συνεχίσει και να κλιμακώσει τις επιθέσεις της απέναντι στους γειτονές της ή με υβριδικές ε, επιθέσεις στις κοινωνίες σας ο αγώνας για τη δημοκρατία σε κάθε χώρα είναι δικαίωμα κάθε χώρας. Κάθε έθνος έχει δικαίωμα στη δημοκρατία και εμείς θα συνεχίσουμε να αγωνιζόμαστε για να προστατεύουμε τη χώρα μας υπέρ της χώρας μας, αλλά μην ξεχνάτε ότι είμαστε στο μέτωπο εμείς και με αυτόν τον τρόπο βοηθούμε τις δικές σας κοινωνίες, τους πολιτικούς σας, τις κυβερνήσεις σας, να αποφασίσουν πώς θα δράσουν αποτελεσματικά, προκειμένου να διατηρηθεί δικιά σας ευημερία, η δικιά σας η ασφάλεια και πώς θα συνεχίσετε στο δρόμο αυτό της ανάπτυξης που ακολουθείτε τα τελευταία 70 παραπάνω χρόνια μετά από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ πολύ. Διστάζω να πιέσω να πάρει το λόγο, αλλά συνάδελφοι, για το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Η Ουκρανία είναι θύμα όχι μόνο της επίθεσης της Ρωσίας, αλλά και της δικής μας ίσως ασυναρτησίας και μη συνοχής. Μιλήσατε για την προσάρτηση της Κρυμαίας. Ποια ήταν η ανταπόκριση εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σημαντική. Αλλά η Ρωσία βλέπει τι γίνεται πολλές φορές με τη στάση κάποιων σε... Αν δείτε για κάποια θέματα. Στο Ισραήλ τα σύνορα είναι του Ισραήλ είναι αυτά του 47, μετά του 65. Ε, δεχθήκαμε αυτό το οποίο γίνεται στο υψίπεδο του Γκολάν, στην, ε, στα Ιεροσόλυμα. Ε, έχουμε εξαιρετικές σχέσεις με το Ισραήλ, παρά το γεγονός ότι κάνει πράγματα αρνητικά. Το ίδιο κάνει με τη Ρωσία, που κάνει για παράδειγμα με την Ουκρανία. Δεν έχουμε λοιπόν συνεκτική ε, πολιτική. Έχουμε λοιπόν να κάνουμε στην Δύση με το κουτί της Πανδώρας. Τι γίνεται. Στον Αγκόρνο Καραμπάχ οι συμφωνίες τι λένε. Ότι το τελευταίο σημείο μετά που αναφέρει την ε, ε, δαφική κυριαρχία των Αγκόρνο Καραμπάχ μιλάμε για τα κυρίαρχα δικαιώματα των πολιτών της. Δίπλα έχουμε το πρόβλημα της Οσετίας. Καταλαβαίνετε λοιπόν πώς αυτή η ασυνέπεια η δική μας με απασχολεί για αυτό που συμβαίνει σε αυτές τις περιπτώσεις και αυτό με αυτό υποφελείται η Ρωσία και στείνει σενάρια παρεμφερή. Το ερώτημά μου στις ε, συμφωνίες του Μίνσκ και της Μαδρίτης όπου η Ρωσία και οι δυτικές δυνάμεις συμφωνούν τι έχουμε, ε, τι σημαίνει για τους κατοίκους της Οσετίας και ποιος είναι ο παραλληλισμός ε, με την κατάσταση στην Κρυμαία. Επίσης, μιλήσατε για τις ε, συμφωνίες της ε, Ράδα, της Ουκρανία. Λέτε ότι δεν επηρεάζει τις συμφωνίες του ΜΙΚ. Βεβαίως, διότι έτσι δίδεται η δυνατότητα στην δική σας ε, την Προεδρία να δράσει και δεν μπορεί. Στο σημείο 4 της Συμφωνίας του ΜΙΣΚ αναφέρεται ότι ε, στο Λουχάνς και στο Ντονέσκ βλέπουμε να υπάρχει βούληση αυτόνομης διακυβέρνησης. Πότε θα εφαρμοστούν με πιστότητα όλες αυτές οι, οι, όλη η δεύτερη συμφωνία του ΜΙΣΚ και κυρίως τα σημεία 4 και 11. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπουστινάρου. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρία Υπουργέ, κύριε Πρέσβη, θα πρέπει να σας πω ότι είναι εντελώς άδικα να λέγεται ότι φτάνει τα θύματα διότι κάποιο τους επιτέθηκε. Δεν θα πρέπει κανεί να το λέει, ούτε εδώ ούτε στο κοινοβούλιο, διότι υπάρχει σαφής διαφοροποίηση. Ο, ε, αυτός που επιτίθεται είναι αυτός ο οποίος ε, φέρει την ευθύνη διότι καταστρατηγεί το διεθνές δικαίο και όχι το θύμα. Θέλω να γίνει αυτό απόλυτα σαφές, διότι στην περίπτωση της Καταλωνίας εγώ ήμουν υπέρ της ε, ενότητας και της ε, ενότητα της ρευστής σε όλη την Ισπανία. Γιατί ο διεθνές δίκαιο δεν εφαρμόζεται εδώ στην ε, Ουκρανία και εδώ έχουμε εισβολή. Γιατί δεν ε, υπάρχει η απόδοση ευθύνης στον αυτόν που επιτίθεται και καταστρατηγεί το διεθνές δίκαιο. Δεν μπορούμε να είμαστε επιλεκτικοί σε μία περίπτωση να λέμε ότι ναι, ε, σεβόμεθα ότι έγινε, στην άλλη το ανεχόμαστε, το δεχόμαστε. Συμφωνώ απόλυτα λοιπόν μαζί σας και με τη θέση της χώρας σας, διότι αγωνίζεστε για να διασφαλίσετε την εδαφική σας ε, ακαιρεότητα και αυτό δεν είναι κάτι το οποίο διαπραγματεύεται μια χώρα. Μια χώρα στην οποία κάποιος άλλη χώρα επιτίθεται έχει δικαιώματα και υποχρεώσεις που του παρέχει το διεθνές δίκαιο, δηλαδή το δικαίωμα πρωτοπόρο να προασπιστεί τα συμφέροντά του και την εδαφική του ακυριότητα. Έχω ένα ερώτημα. Μου είπαν πρόσφατα ότι κάποιες ρωσικές μονάδες προετοιμάζουν τρομοκρατικές επιθέσεις, επιθέσεις συγγνώμη, σε εγκαταστάσεις ε, ρουμανικές στην Ουκρανία. Είναι αληθές αυτό? Μπορείτε να μας εξηγήσετε αυτή την ε, νέα διάσταση του υβριδικού πολέμου που χρησιμοποιεί τις μειονότητες στην Ουκρανία ή για να αποδυναμώσει ακόμη περισσότερο τη συνοχή του κράτους ή για να, με τα, να τα να τη θυματοποιήσει και για να δημιουργήσει προβλήματα μεταξύ άλλων γειτόνων μεταξύ τους. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Δεν βλέπω να ζητά κανείς άλλο το λόγο. Όχι. Πιστεύω ότι ο κύριος Μποστενάρου δεν κατάλαβε τι ακριβώς είπα. Πολύ σύντομα. Συμφωνεί μου κύριε Μποστενάρου, και εσείς και εγώ. Εγώ είμαι υπέρ της δαφικής ακεραιότητας της Ουκρανίας, της Συμφωνίας Βουδαπέστης και λέω ότι η Ουκρανία υπέστη επίθεση. Αυτό το οποίο θέλω να τονίσω είναι της δικαίη μας ε, ε, ασυνέπεια κατά κάποιο τρόπο. Και δεν θα πρέπει μόνο να ψέγουμε για την κακία του τον εισβολέα, αλλά και εμείς ώρες-ώρες ε, ε, πρέπει να δούμε πώς ακριβώς έχουμε ενεργήσει σε τέτοιου είδους περιστάσεις και ποια ήταν η στάση μας. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα θα ήθελα να υπενθυμίσω ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο λαμβάνει υπόψη τα θέματα τα αυτά της Ουκρανίας, της Κρυμαίας, τα εξετάζει, τα παρακολουθεί. Έχουμε πολλοί άριθμα ψηφίσματα που εγκρίθηκαν με πολύ μεγάλη πλειοψηφία υπέρ εκ μέρους των μελών της, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ό,τι συμβαίνει με τις καταστρατηγήσεις, παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, τα θύματα στην Ουκρανία, τα δικαιώματα των ε, μειονοτήτων. Το λαμβάνουμε υπόψη. Θα ήθελα να σας μιλήσω για κυρώσεις. Βεβαίως θέλουμε να διατηρηθούν οι κυρώσεις, αλλά ζητήθηκαν οι κυρώσεις να επιβληθούν για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. Και το συζητούμε αυτό, να ξεπεράσει το χρόνο. Αυτό είναι ένα θέμα το οποίο συζητούμε, αλλά μήπως αυτό κατά κάποιο τρόπο αποδυναμώνει την ενότητα. Δεύτερον, ποια είναι τα κύρια εμπόδια κατά την άποψή σας ε, για την δημιουργία και την αποστολή αυτής της ερηνευτικής δύναμης του ΟΗΕ. Τι θα μπορούσαμε εμείς ως Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να αναλάβουμε ως πρωτοβουλία για το θέμα αυτό, λαμβάνοντας υπόψη την ε, πρώτη επέτειο της ε, παράνομης προσάρτησης της Κρυμαίας. Ευχαριστώ κυρία Φωτίγα και ευχαριστώ πολύ που σε φυστάτε την προσοχή σε αυτό το γεγονός των Τατάρων της Κρυμαίας και της παράνομης προσάρτησης της. Γνωρίζετε ότι αυτά τα θέματα μας απασχολούν πάρα πολύ και ξέρουμε ότι τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ενδιαφέρονται και τα μέλη της δικής σας Επιτροπής. Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις σας. Θα προσπαθήσω να απαντήσω. Πρώτον, σε ό,τι αφορά τα ειδικά πολιτικά χαρακτηριστικά της συμφωνίας των συμφωνιών του Μίνσκ. Είναι δύσκολο να προχωρήσει κανείς και να κάνει κάποια πρόοδο και να βρει ε, προθυμότητα από την κοινωνία για τα πολιτικά θέματα ε, της συμφωνίας του Μίνσκ στο βαθμό που δεν έχουμε επιλύσει το θέμα της ασφάλειας επιτόπου. Καθημερινά σκοτώνονται ή τραυματίζονται ε, στρατιώτες και άμαχος πληθυσμός μας. Καταστρέφεται υποδομή. Κάθε μέρα που περνάει, όσο έχουμε αυτές τις ομές και βίες επιθέσεις ε, στον άμαχο πληθυσμό και ε, σε εκείνους που υπερασπίζονται τη χώρα μας. Δεν γίνεται αυτό. Ό,τι μπορούσαμε κάναμε και ακόμα περισσότερο. Ήδη έχουμε ανταποκριθεί στο πολιτικό σκέλος των συμφωνιών του Μίνσκ. Ιδιαίτερα σε σχέση με αυτό που αναφέρεται για την περιφέρεια του ε, Ροχάνσκ και του Ντονιέτσκ. Έχουμε ειδικό νόμο που εγκρίθηκε από τη Ράντα, τη Βουλή μας, εξέπνευσε το Σεπτέμβριο του 2017, ε, αλλά παρατάθηκε από την ε, Ουκρανική Ράντα. Δηλαδή, το Κοινοβούλιο μας λαμβάνει πολύ σοβαρά υπόψη, όσο και υπεύθυνα την προσήλωσή μας και τη δέσμευσή μας. Ε, όσο δύσκολες και να είναι οι συμφωνίες και οι λύσεις που προτείνονται στις συμφωνίες του Μίνσκ όσον αφορά την κοινή και ενωμένη αντίδραση στις διάφορες προκλήσεις που από κοινού αντιμετωπίζουμε. Και προφανώς ε, η Ουκρανία είναι μία και μόνο από τις αιστείες τις φλεγόμενες που πρέπει αυτή τη στιγμή να αντιμετωπίσουμε την εισβολή και την επιθετικότητα της Ρωσίας. Κοιτάξτε, θα πρέπει να θυμόμαστε ότι δυστυχώς η δική μας αδύναμη κοινή αντίδραση σε προηγουμένες δράσεις της Ρωσίας επέτρεψαν στη Ρωσία ακριβώς ε, να ε, αυξήσει τις ορέξεις ε, και τις επιβουλές της. Εάν το 2008, για παράδειγμα, ήμασταν πιο συντονισμένοι και πιο σοβαρά αντιδρούσαμε στην επίθεση στη Γεωργία, και η Ουκρανία μέσα. Δεν βγάζω την Ουκρανία απ' έξω, ούτε ρίχνω το φταίξιμο σε χώρε ΝΑΤΟ ή τη Ευρωπαϊκή Ένωση ή μόνο τι δυτικέ χώρε, σε καμία περίπτωση. Και εμεί στην Ουκρανία δεν αντιδράσαμε αρκετά στεναρά και αποτελεσματικά και δεν κρούσαμε τον κόδωνα του κινδύνου όταν επιτέθηκε η Ρωσική Ομοσπονδία στη Γεωργία και επιτρέψαμε τις ρωσικές ε, ρέξεις και επιβουλές να αυξηθούν, γιατί Πούτιν ότι υπάρχει ατιμορρησία από τη Δύση. Παρόλο που χαρήκαμε πολύ από τις αρχικές ε, κυρώσεις σχετικά με την παράνομη προσάρτηση της ε, Κρυμαίας, θα σας το πω έξω από τα δόντια. Νομίζω ότι οι κυρώσεις αυτές ήταν πολύ ασθενείς και επέτρεψαν ακριβώς τον Πούτιν να του ανοίξει η όρεξη και να προχωρήσει στην επιθετικότητα και να, και να επιτεθεί στην ε, Ανατολική Ουκρανία. Άρα, είναι περίπλοκα αυτά τα θέματα και ταραγμένες διάφορες αιστείες ανάφλεξης ε, που θα πρέπει να πάρουμε υπόψη μας και συμφωνώ απολύτως με αυτά που είπατε ε, ότι θα πρέπει να προσιλωθούμε ε, το διεθνές δίκαιο. Αυτό είναι το κράτος δικαίου. Αυτό το δίκαιο μας επέτρεψε να ζήσουμε και να αναπτυχθούμε και να εξυγχρονιστούμε και να ενισχυθούμε όλα αυτά τα χρόνια μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Συμφωνήσαμε για ένα διεθνές δίκαιο και ένα πλαίσιο. Εμείς βάλαμε τους κανόνες για μας τους ίδιους και σε μας εναπόκειται πάντα να τους στηρούμε τους κανόνες αυτούς και στο γράμμα τους και να μην βρίσκουμε προφάσεις για να δικαιολογούμε κάποιους και κάποιους άλλους να τους αφήνουμε να αποκλείουν και να αφίστανται από το γράμμα του νόμου σε άλλες περιπτώσεις. Για τις κυρώσεις λοιπόν, και θα επανέλθω στις ερωτήσεις σας, έχω να πω το εξής. Πολλές φωνές ακούμε και πολλές φορές ευρωπαϊκές πρωτεύουσες που ενδιαφέρονται να έχουν κάποιο είδους χαλάρωση των κυρώσεων, ε, προοδευτικά. Αυτή η συζήτηση είναι τελείως αντιπαραγωγική. Αυτό θέλει να κάνει η Ρωσία. Να δημιουργήσει τριβές και χάσμα και να βάλει σφήνα ανάμεσα στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Και ψάχνει το πιο αδύναμο κρίκο, το θυμάστε αυτό το βρετανικό τηλεπαιχνίδι, το πιο αδύναμο κρίκο για να του επιτεθεί και να μας αποδυναμώσει. Και να σπάσει αυτή την ενότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη Διατλαντική. Ισχυροί είσαστε μόνο όταν είστε ενωμένοι και ικανοί είστε όταν είστε ενωμένοι. Και αυτή είναι όλη η κεντρική ιδέα, ότι, στην οποία οικοδομήθηκε η ίδια Ευρωπαϊκή Ένωση και βασίζεται. Άρα έχει σημασία να διαφυλαχθεί αυτή η ενότητα. Ούτε θέλουμε εμείς στην Ουκρανία να δούμε να συνεχίζονται αυτές οι αντιπαραγωγικές συζητήσεις κάθε εξάμεινο για το εάν και κατά πόσο θα πρέπει να αρθούν ή όχι οι κυρώσεις. Αν δεν υπάρχει καμία προθυμία από την άλλη πλευρά τη Ρωσική να σταματήσει την επιθετική της συμπεριφορά προς την Ουκρανία. Η μία δυνατότητα είναι να επεκταθούν ε, και να παραταθούν οι ε, κυρώσεις για ένα χρόνο αντί για το εξάμεινο και το άλλο είναι να ενταθούν οι κυρώσεις. Δεν ισχύει το επιχείρημα ότι δεν αποδίδουν. Δεν θα είχε τέτοια δυσφορία απέναντι σε αυτές η Ρωσία ε, αν δεν απέδιδαν. Και δεν μπορούμε να καθίσουμε να περιμένουμε δεήσει η Ρωσική Ομοσπονδία να σεβαστεί το διεθνές δίκαιο. Βλέπω και στον τύπο κάποια δημοσιεύματα. που λέγουν ότι μάλλον προετοιμάζουν επιθέσεις κατά της ρωμανικής κοινότητας στην Ουκρανία. Αποδείξεις δεν έχω τέτοιες, οπότε δεν θα ήμουν σε θέση να το επιβεβαιώσω αυτό. Παρόλα αυτά, Σήμερα ακριβώς στην Ουκρανία στην Υπερκαρπαθία είχαμε μια επίθεση εκεί ε, στα ουγγρικά γραφεία της κοινότητας εκεί πέρα από τα Καρπάθια. Ε, είναι η δεύτερη επίθεση αυτό το μήνα στους Ούγγρους. Καθώς γίνεται συζήτηση για την στην Ουγγαρία σε σχέση με ένα νόμο εκπαιδευτικό πάρα πολύ προεδευτικό και ρίξει και έλευθο, όπου αντιμετωπίζουμε και το θέμα ε, της διδασκαλίας ε, στη μητρική γλώσσα. Γίνεται μια συζήτηση λοιπόν Ουκρανίας, ε, ε Ουγγαρίας ε, συναισθηματικά φορτισμένη και έντονη και ακριβώς αυτή τη χρονική στιγμή είδαμε δύο επιθέσεις κατά της, γραφείο γραφείων της Ουγγρικής κοινότητας. Η δική μου οικογένεια κατάγεται από την περιοχή αυτή, όπου ανέκαθεν υπήρχαν διαφορετικές εθνοτικές ομάδες και μειονότητες που ε, συνεβίωναν ε, αρμονικά. Και με πίστη, λέει ο κύριος Μποστινάρου, και με πίστη και με σεβασμό, βεβαίως. Εγώ δεν μεγάλωσα εκεί και παρόλο που είμαι Ουκρανή και πήγαινα μόνο το καλοκαίρι ε, και, να δω τη γιαγιά μου, ε, μιλώ Ουγγρικά ε, για να μπορώ να μιλάω με το γείτονα και να το χαιρετάω και να τους λέω καλημέρα, καλησπέρα, τι κάνετε, να σέβομαι τις θρησκευτικέ τους και άλλες εορτές και ε, τούμπαλιν. Ποτέ λοιπόν δεν υπήρχαν ε, εντάσεις, τριβές ή επιθέσεις σε Ουκρανούς και σε Ούγγρους. Η αστυνομία έχει πάει εκεί και διερευνά την υπόθεση ήδη και ελπίζω να βρεθούν οι ένοχοι και να προσαχθούν στη δικαιοσύνη. Αλλά αυτές οι προκλήσεις δεν είναι εσωτερικού τύπου, είναι ορμόμενες από κάποια μέρη πολύ μακριά από τα δικά μας σύνορα. Και είχαμε και στο παρελθόν με την Πολωνία ε, κάποια προβλήματα και για πρώτη φορά στα 25 χρόνια της ανεξαρτησίας υπήρξε επίθεση σε πολωνικό προξενείο στην Ουκρανία. Αυτά είναι ξένης κοπής και έμπνευση. Δεν είναι ντόπια φαινόμενα. Και ε, αυτοί που τα κάνουν δεν ενδιαφέρουν να ευημερεί η κοινωνία στην Ουκρανία ούτε να πάει μπροστά το κράτος. Πραγματικά ήθελα να το τονίσω. Νομίζω ότι απάντησα στις ερωτήσεις σας πάνω κάτω. Ε, καλώς, δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλοι συνάδελφοι που να θέλουν το λόγο για σχόλια ή ερωτήσεις. that, uh, Νομίζω ότι εδώ μπορούμε να ολοκληρώσουμε τη σημερινή μας συζήτηση. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύρια που ήρθατε. Παρακαλώ να χειροκροτήσουμε μαζί την ε, ε, εξαιρετική προσκεκλημένη. Thank you. Thank you very much. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνάδελφοι, θα πρέπει να κλείσουμε τη συνεδρίαση αυτή. Στα διάφορα έχει να προσθέσει κανείς κάτι. Εάν δεν υπάρχουν λοιπόν παρατηρήσεις, θα ήθελα να αναφέρω ότι η επόμενη συνεδρίασή μας είναι στις 21 και 22 Μαρτίου. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τη συμμετοχή τους στη σημερινή συνεδρίαση, τους διερμηνείς για την εργασία τους και οι διερμηνείς ευχαριστούν την Πρόεδρο και την Γραμματεία την συμμετοχή. Σας ευχαριστώ πολύ όλους.